Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε την απογευματινή συνεδρίαση με το σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη που έχει να κάνει με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της δικαιοσύνης ε, ε, και των ιστορικών υποθέσεων. Έχουμε το Φαμπρίζ Λετζέρι ε, από τη Frontex και την παρουσίαση της αξιολόγησης τροτότητας εξαμηνία έκθεση 1 του 2019. Γνωρίζετε ότι στην προηγούμενη θητεία ένα από τα βασικά θέματα της δικής μας Επιτροπής ήταν και τα θέματα που ε, είχαν να κάνουν με ε, τη Frontex, που είναι η ε, Ευρωπαϊκή Συνεροφυλακή και Ακτοφυλακή. Το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή ΛΥΒΕ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, εξασφάλισε τη δυνατότητα λειτουργίας του Frontex Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα θεσμικά όργανα ολοκληρώνουν τον τελευταίο γύρο της νομοθετικής ε, διαδικασίας ε, για το Frontex ε, με τη διόρθωση των σφαλμάτων. Ελπίζουμε ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ στα τέλη του έτους. Συνεχίζουμε τις επαφές μας με τους οργανισμούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνη και στα πλαίσια αυτά θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Φαμπρίς Λεζερή, εκτελεστικό διευθυντή του Frontex, που θα μα παρουσιάσει τα καθήκοντα και τι δραστηριότητε, καθώ επίση και ε, την εξαμηνία έκθεση, την πρώτη του 2019, για την αξιολόγηση της τροτότητας. Έχετε το λόγο για 20 λεπτά το πολύ. Καλώς ορίσατε. Thank you very much, uh, Madam Chair. Honorable... Αξιότιμη Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή, η επανεκλογή σας και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δυνατότητα που μου δίνεται να σας παρουσιάσω σήμερα τις δραστηριότητες ε, της ε, Frontex της Ευρωπαϊκής Συνοριακής και Ακτοφυλακής Πρώτα απ' όλα όμως, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας πω και τι κάνουμε στα πλαίσια της φυστάμενης εντολής μας, αλλά και στο πλαίσιο της ε, εκπόνησης της νέας εντολής ε, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη του έτους. Ποιο είναι το DNA του οργανισμού μας. Μπορεί να διερωτηθείτε γιατί να υπάρχει η Frontex, η Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Εκτοφυλακή. Η απάντηση που έχω να σας δώσω είναι πολύ απλή. Χρειάζεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει τον χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης ε, και ασφάλειας ε, και γι' αυτό θα πρέπει τα εξωτερικά μας σύνορα να λειτουργούν σωστά. Που σημαίνει ότι στις δραστηριότητες μας ε, θα πρέπει τα εξωτερικά σύνορα να μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που άπτονται της ε, παράτυπης μετανάστευσης και όχι μόνο βέβαια, το διασυνορικό έγκλημα στα εξωτερικά σύνορα, όπως και πρόληψη της τρομοκρατίας. Μακροπρόθεσμα δε, θα πρέπει να μπορούμε να αναπτύξουμε και εναρμονισμένες ε, δυνατότητες και τεχνολογίες για να φροντίσουμε τα 750.000 νόμιμους ε, ταξιδιώτες. 750 εκατομμύρια, συγγνώμη. Είχα ξαναπάει την 1η Απριλίου σε μια κοινή συνεδρίαση με άλλες επιτροπές και θέλω να επαναλάβω τώρα σε δική σας την Επιτροπή ακριβώς επειδή διαβρύνεται η εντολή και στελεχώνεται με περισσότερα μέσα η Frontex, τελεστικός διευθυντής στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρέπει να παρίσταται για σκοπούς λογοδοσίας. Θα ήθελα να σας πω τώρα δύο πράγματα για τις στρατηγικές δραστηριότητες, όπως είναι εκτίμηση τροτότητας και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων δημιουργίας υποδομών και δυνατοτήτων. Και μετά θα περάσω σε κάποια στοιχεία για την εφαρμογή της μελλοντική μας εντολής, την εκτέλεση της εντολής μας σε στρατηγικό έργο της Frontex. Πώς μπορεί να ανακεφαλωθεί σε, με λίγα λόγια. Είναι τεχνη... Είναι η στρατηγική της ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που το ενέκρινε το Δικτικό Συμβούλιο φέτος την Άνοιξη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται και στη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και φυσικά και του Ευρωκοινοβουλίου που διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά το πολιτικό πλαίσιο. της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης συνόρων. Δεν αφορά αυτό όμως μόνο τι κάνει η οργάνωσή μας, αλλά είναι και ένα κοινό πλαίσιο για τις εθνικές αρχές, που είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο συνεισφέρουν στη διαχείριση των συνόρων, όπω είναι η ακτοφυλακή και οι δραστηριότητε, ε, αυτέ, βέβαια όσο σχετίζονται με την φύλαξη των συνόρων. Υπάρχει και ένα άλλο στρατηγικό στρώμα, ένα άλλο στρατηγικό επίπεδο που είναι η ψυχολογική στρατότητα. Αναφερθήκατε σε αυτό κυρία Πρόεδρε. Αυτή η δραστηριότητα πρωτοξεκίνησε το 2017 με βάση τον προηγούμενο κανονισμό που είχε κριθεί και τεθεί σε ισχύ το 2016. Τώρα Πρόκειται για μια συστηματική αξιολόγηση που διενεργεί η Frontex ό,τι αφορά τις δυνατότητες διαχείρισης εξωτερικών συνόρων όλων των κρατών μελών. Γίνεται λοιπόν σε αιτήσια βάση και τώρα είναι σε εξέλιξη ο τρίτος κύκλος αξιολόγηση. Θα μπορούσα να το συγκρίνω με ένα check-up ιατρικό αυτό που κάνουμε. Βασιζόμαστε σε στοιχεία που μας παρέχουν ε, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών Έχουμε μία κοινώς ε, συμπεφωνημένη μεθοδολογία και κάποιους δείκτες ε, κοινούς για, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν επί το, ώστε να εφαρμόζεται ο κώδικας ε, Σέγγεν και να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση ε, γίνεται με επαρκή φόρου και μέσα και ότι υπάρχει επαρκή ευελιξία για την αντιμετώπιση αναδειωμένων απειλών. Τον Ιούνιο, το Ευρωκοινοβούλιο, όπως κάθε χρονιά, όπως πάντοτε, τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν την έκθεση παραγμένων του οργανισμού, την ενημέρωσή μας επίσης ε, για τα βασικά πορίσματα και ευρήματα. Βεβαίως ως ευρωβουλευτές μπορείτε να συναγάγετε τα δικά σας συμπεράσματα, όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο νομοθέτης, ο συνομοθέτης να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται ορισμένε φορές σωστά η νομοθεσία. Σύντομα επακολουθεί η δεύτερη έκθεση. Την αναμένουμε περίπου για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Και θα την λάβετε κι εσείς βέβαια. Τότε θα την έχουμε έτοιμη. Υπάρχουν προκλήσεις ε, για συστηματικούς ελέγχους στα σύνορα. Ήδη τις ε, προκλήσεις αυτές τις είχαμε εντοπίσει και βλέπουμε να επιμένουν ιδίως όταν είναι υποχρεωτική αυτή η έλεγχη ε, σε σχετικές βάσεις δεδομένων. Μιλάω για το ΣΥΣ, το ΒΙΣ, και όχι μόνο για ελέγχους σε επικός τρίτων κρατών, για ταξιδιώτες μιλάω. Και ξέρετε, όποιος εισέρχεται ή ξέρχεται του χώρου Σέγγεν θα πρέπει να ελέγχεται. Να αντιπαραβάλλεται τα στοιχεία του με αυτά που περιλαμβάνει το ΣΥΣ, το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν. Και όλα αυτά οξύνονται από το γεγονός πως υπάρχει ε, σημαντικό έλλειμμα προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ορισμένες εθνικές υπηρεσίες δεν έχουν επαρκές προσωπικό για διαφόρους λόγους στην κάθε περίπτωση. Όμως, ο εκτιμόμενος αριθμός προσωπικού που λείπει είναι πάνω από 5.000 για φέτος και πρόκειται για μια πολύ ε, ευαίσθητη δραστηριότητα, όπως καταλαβαίνετε. Πολλά κράτη-μέλη θεωρούν πως ποτέ αυτό είναι ένα είδος ε, check-up έχει δηλαδή να κάνει με πολύ ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι υπάρχει και ανάγκη για διαφάνεια ε, στην έκθεση αυτή. Γιατί μέσω των θεσμικών οργάνων και ιδίως του Κοινοβουλίου φτάνει και στους πολίτες αυτή η ενημέρωση. Ιδίω εν ώψη των ε, μελλοντικών εξελίξεων, καθότι θα τεθεί σε ισχύ ο νέο κανονισμό, ε, βεβαίω και είμαι στη διάθεσή σα στην Επιτροπή σα ε, στο Κοινοβούλιο γενικώ να έρθω και να σα πω πώ μπορούμε να βρούμε τρόπου για να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία, χωρί να διακινδυνεύσουμε τι σχέσει μα με τι εθνικέ αρχέ που εδράζονται στην εμπιστοσύνη. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα με την Επιτροπή σα, Αν με επιτρέπετε να αναφέρω και κάποιε δραστηριότητε ε, ανάπτυξη επιχειρήσεων και δυνατοτήτων. Όσοι γνωρίζετε τον οργανισμό μα, ήδη τα ξέρετε αυτά, αλλά να σα πω, πως αυτή τη στιγμή έχουμε μεταξύ 1.300 και 1.500 ε, συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες που αναπτύσσονται ε, στο πλαίσιο των διαφόρων ε, επιχείρησεων ο ειδών Θέμης, και Μινέρβα. Πρώτη στην Ελλάδα, δεύτερη στην Ιταλία, τρίτη στην Ισπανία και θα έχουν και στην Αλβανία σύντομα μια επιχείρηση και κάποιε άλλε δραστηριότητε σε διάφορα χερσαία σύνορα και σε διάφορα αεροδρόμια. Θέλουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Ε, παρακολουθούμε 24 ώρου βάσεως ε, και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Έχουμε ενισχύσει, στελεχώσει καλύτερα ε, τα κέντρα ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επιτηρούμε και να έχουμε καλύτερη εικόνα των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σέγγιν ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενισχύουμε επίσης την ανάλυση κινδύνου να σας δώσω ένα παράδειγμα συνεργασίας που έχουμε. Πριν από κάποιους μήνες μαζί με την ΕΑΣΟ και την Europol κάναμε μία έρευνα για τις ε, παράτυπες ε, δευτερογενείς μετακινήσεις. Δευτερογενείς μετακινήσεις, τι θα πει αυτό. Ε, αν θέλουμε να λειτουργεί και να το αντιλαμβάνεται έτσι ο κόσμος, ότι λειτουργεί ο χώρος του Σέγγεν, ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Όπως είπα, θα αναπτύξουμε μια επιχείρηση στην επιχείρηση στην Αλβανία. Συμφωνήσαμε με τη χώρα αυτή μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει επικυρώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αποστολή στα χέρια σύνορα μεταξύ Ελλάδα και Αλβανία, αλλά από την αλβανική πλευρά τη Μεθορίου ε, θα αναπτυχθεί αυτή η επιχείρηση για τον έλεγχο και τη διατήρηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, αλλά και την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματο. Και επίση έχει στόχο ευρύτερα τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, έχοντα υπόψη το γεγονό ότι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων είναι αντικείμενο μια ιδιαίτερη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικών Βαλκανίων. Συνοριαφύλακε τώρα, εν γέννη, έχουν ένα σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας. Εδώ μιλώ για την πρόληψη, την οντοπισμό διεθνών εγκληματιών και πρόληψη της τρομοκρατίας. Θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, γι' αυτό άλλωστε συνεισφέρουμε και στη καλή λειτουργία των εξωτερικών συνόρων, που σημαίνει ότι αυτά τα εξωτερικά σύνορα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ένα φίλτρο, ώστε ακόμη και απειλέ για την ασφάλεια να ε, γίνονται αντιλητές, να εντοπίζονται μεγάλο επιτεύγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός ότι επειδή δεν έχουμε τους νομικούς πυλώνες που είχαμε πριν, μπορούμε τουλάχιστον έτσι να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, να έχουμε λιγότερα στεγανά και αυτό το έκανε και τα τελευταία χρόνια η Frontex ενισχύοντας και αναπτύσσοντας τη δραστηριότητα στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας με ξεκάθαρη και ενισχυμένη συνεργασία με τη Europol φυσικά με τις Εθνικές Αρχές Επιβολής του Νόμου, τελωνιακούς, αστυνομικούς και τώρα με βάση την εντολή μας θέλουμε και με τη Eurojust ε, καλύτερη συνεργασία και με τις αποστολές και ΠΑ. Χάρη στην ενισχυμένη εντολή μας ότι αφορά τη χρήση, συλλογή χρήση και επεξεργασία και ανταλλαγή με προσωπικού χαρακτήρα, θα είμαστε τα αυτιά και τα μάτια, όπως λέμε μερικές φορές, ε, ε, των αρχών επιβολής του νόμου. Όμως αυτά όλα τα στοιχεία τα ανταλλάσσουμε ουσιαστικά με τις αρμόδιες αρχές που κάνουν τη δουλειά επιτόπου, που προχωρούν στις έρευνες και στους ελέγχους. Και στο τμήμα τη ακτοφυλακή με το με διάφορους άλλους φορείς για την αλία, για την προστασία της θάλασσας. Το 2016 έχουμε κοινέ εντολές ε, για κοινή ανάπτυξη κάποιων ε, επιχειρήσεων ακτοφυλακής. Παραδείγματο χάρη, εντοπίζουμε πετρελοκυλίδες ε, ή άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές ή ε, παράνομη αλία, δαστέρες παράνομης αλίας. Βέβαια, διάσωση, έρευνα και διάσωση είναι το βασικό ίσως, για εσάς τουλάχιστον. Και θέλουμε να έχουμε περισσότερες ναυτικές δυνατότητες, θαλάσσιες δυνατότητες για να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες ε, των ε, αρχών ε, που συντονίζουν τις υπηρεσίες της επιχειρήσης έρευνας και διάσωσης. Και άρα έχουμε βελτιώσει τη δράση μας στον τομέα αυτός, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα. Προς το παρόν η Ιταλία, η Ισπανία. Δύο και τέσσερις Οκτωβρίου θα γίνει μια συγκεκριμένη συνδοσιά τη επιχειρήση επιχειρήσει ε, και διάσωση 2 και 3 Οκτωβρίου. Έχω ήδη ενημερώσει την Επιτροπή σα. Θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για την ε, εφαρμογή του κανονισμού τη ε, Frontex. Αλλά βεβαίω θα συμμετέχουμε έστω με γραπτή συνεισφορά. Αν δοθεί δε δυνατότητα να γίνει κάπω αλλιώ, ε, να έχουμε μια άλλη συμμετοχή. Θα δούμε υλικοτεχνικά πώ μπορούμε να το οργανώσουμε. Απλά σα το λέω, 2 και 3 Οκτωβρίου ο πρόεδρο του ΔΣ έχει οργανώσει αυτή τη στρατηγική διάσκεψη, σύνοδο. Τώρα, να σα κάνω μια παρουσίαση συνοπτική των δραστηριότητων για τις επιστροφές. Στο πλαίσιο τη διαχείριση τη παράτησης μετανάστευση. Ήδη έχουμε ενισχύσει την εντολή μας από το 2016 επ' αυτού. Η δική μας συμβολή είναι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, εθνικές αρχές, γιατί αυτοί κάνουν, ε, λαμβάνουν τις αποφάσεις, δεν μπορούμε εμείς ε, για τις επιστροφές να πάρουμε κάποια απόφαση. Τι κάνουμε όμως εμείς, ε, βοηθάμε στον εντοπισμό, στην ταυτοποίηση, στη μεταφορά των ατόμων αυτών είτε με μισθωμένες ναυλωμένες πτήσεις ή με τις τακτικές ε, πτήσεις. Το 19 επιστρέψαμε γύρω στους 10.000 άτομα σε χώρες ε, τρίτες εκτός Ένωσης. Επίσης, αναπτύσσουμε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και με την ΕΑΖΟ πάνω σε αυτό, γιατί μετά από μια αρνητική απόφαση για την παροχή ασύλου για την παροχή της προστασίας θα πρέπει οι αρχές να είναι σε θέση να ε, εκτελούν τις αποφάσεις αυτές για επιστροφή των ελόγω ατόμων. Συμμετέχουμε επίσης στις προετοιμασίες των μεθοριακών σημείων ελέγχου για το, με το Ιουλίζα e θέλουμε να εφαρμοστεί στο το σύστημα ε, σοδού εισόδων εξόδων και για το αίτιας επίσης και η Frontex θα οργανώσει μια σχετική ενημέρωση. Και έρχομαι στο μέλλον. Ανάπτυξη της νέας εντολής. Η η οποία θα οδηγήσει σε μια βαθιά οργανωτική μετάλλαξη του οργανισμού μας, που έχει ξεκινήσει εδώ και, μια τριετία. Βεβαίως, με το μόνιμο ευρωπαϊκό αυτό σώμα θα ξεκινήσουμε από άλλη πλέον βάση. Τίποτα παρόμοιο δεν υπάρχει μέχρι στιγμή στην Ένωση. Άρα για πρώτη φορά θα έχουμε φορείς ε, επιβολής του νόμου που θα είναι Ευρωπαίοι, θα φέρουν όπλα ε, και ευρωπαϊκή στολή. Ε, να το έχουν υπόψη μας για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Εγώ βέβαια θα σας αναφέρω και στο μέλλον σε σχέση με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Επίσης, αυτό που αλλάζει πραγματικά τα δεδομένα με τον νέο αυτοκανονισμό είναι το βελληνικές, η κλίμακα των επιπλέον πόρων δεν μιλώ μόνο για τον προπολογισμό αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό. Αλλάζουν τα δεδομένα, όπως είπα. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να ε, φροντίσουμε ότι εμείς αναπτύσσουμε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ε, των κρατών μελών και των εθνικών αρχών. Είναι και θέμα λογοδοσίας, ευθύνη. ώστε και εσείς να είστε σίγουροι, εσείς οι ευρωβουλευτές, ότι αυτό που κάνουμε εμείς και ο τρόπος με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε το δημόσιο χρήμα είναι χρήσιμο και τη χάνει σωστή διαχείριση. Κάτι άλλο που τα δεδομένα βέβαια είναι αυτό το European Standing Core, αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα, το διακίνηση με 10.000 ε, άτομα, κατηγορία 1 που είναι Ευρωπαίοι και κατηγορίες 2 και 3 εθνικοί ε, αξιωματούχοι. Also, ε, develop... Ε, αποσπασμένοι λοιπόν φύλακες και θα έχουμε και κάποια γραφή για την υλικοτεχνική διαχείριση, τα logistics. Γιατί όταν λέμε για 10.000 ε, φύλακες, πρέπει να γίνει αποκεντρωμένη διαχείριση, αν θέλουμε να υπάρχει ευελιξία επιχειρησιακή. Θα ενίσχυσουμε την ανάλυση κινδύνων για περισσότερη πρόληψη με στόχο να μπορούμε να προβλέπουμε, να προ... καταλαμβάνουμε τις εξελίξεις, ώστε να αποφύγουμε και όλες οι δυνατόν να ξεσπούν κάποιες κρίσεις και δεν μιλάω μόνο για παράνομες μεταστατικές ροές, αλλά και μια σειρά άλλη, άλλων απειλών. Πολλές φορές συνδέονται με τρομοκρατία, το έγκλημα ή υβριδικές απειλές ενίοτε. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή, εσωτερικά έχουμε ξεκινήσει προτείνοντας να αναπτυχθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για το επιχειρησιακό μας δόγμα. Με πολύ απλή συλλογιστική. Έχουμε την ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση των εξωτερικό σύνολο. με βάση τρει πυλώνες. Κάθε ένας από αυτούς τους πυλώνες θα είναι ένας από τους τρεις στρατηγικούς στόχους. Ο πρώτος στρατηγικός στόχος είναι η μείωση της τροτότητας των εξωτερικών συνόρων με βάση μια συλλογική ευαισθητοποίηση για την κατάσταση. Δηλαδή, περισσότερη πληροφόρηση για να υπάρχει δυνατότητα πρόληψη, ευαισθητοποίηση, ε, αναγνώριση του τι συμβαίνει. Και τώρα και στο μέλλον. Δεύτερο στρατηγικό στόχο. Ασφαλή και καλά λειτουργούντα Εξωτερικά σύνορα, επιτήρηση σύνορων, αλλά και λειτουργία των σύνοριακών σημείων ελέγχου. Και δεν μιλάμε μόνο για τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές, όπως είπα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια των ταξιδιωτών που ταξιδεύουν νομίμως. Και ο τρίτος στρατηγικός στόχος είναι οι βιώσιμες δυνατότητες ε, ε, ακτοφυλακής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας και ουσύνης ελευθερίας πρέπει να στελεχωθεί με τουλάχιστον 5.000 ε, φυλακέ, για να πω και παραπάνω. Έχουμε έλλειμμα. Θέλουμε τυποποίηση, συντονισμό, περισσότερε νέε τεχνολογίε. Κάποιε φορέ δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιου ε, με τεχνολογία, με κάπου χρειάζεται ε, το ανθρώπινο προσωπικό και κάπου βέβαια μπορεί καλύτερα ένα σύστημα να λειτουργήσει με ένα εξοπλισμό. Αυτό και είναι και ο τρίτος μα στόχο. Τώρα, να αναπτύσσουμε κάποιε υπηρεσίε. Αυτό που θέλουμε να είναι σαφές είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε στα κράτη-μέλη που έχουν και την πρωταρχική ευθύνη. Η διαχείριση συνόρων όμως είναι κοινή ευθύνη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Εμεί είμαστε το επιχειρησιακό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αναπτύξουμε ένα κατάλογο υπηρεσιών ώστε οι εθνικές αρχές, τα κράτη-μέλη να μπορούν βάσει αυτού να καταθέτουν τα αιτήματά τους και να λαμβάνουν σχετική υπηρεσία από τον οργανισμό. Πρέπει να είμαστε και πιο ευέλικτοι. Είναι κάτι που θα το δείτε στο μέλλον στην επιτεροποίηση, σύντομα κιόλα ε, στην επιτεροποίησή σας με την έγκριση ε, του εγγράφου νέου προγραμματισμού, στρατηγικό λοιπόν πλαίσιο, τρεις στρατηγικοί στόχοι, όπως είπα, που θα είναι και η δομή αυτού του ενίου προγραμματισμού. Και θα ολοκληρώσουμε τα εξή. Συμφωνήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα οδικό χάρτη, κοινό χάρτη για την εκτέλεση του νέου κανονισμού και τη δημιουργία αυτού του μόνιμου σώματος. Ήδη έχουμε προετοιμάσει ε, το πρώτο υλικό για την ε, προσλήψεις, ξεκινήσει η διαδικασία σύντομα και το ίδιο σε ό,τι αφορά τα προφίλ. Την περιγραφή εργασίας. Σε ό,τι αφορά τις εθνικές αρχές, έχω οργανώσει πέντε περιφερειακές συνελεύσεις μεταξύ ε, τελών Οκτωβρίου και αρχές Δεκεμβρίου για ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα ανάλυση των επιχειρησιακών προσδοκιών και απαιτήσεων. Αλλά θέλω και να εξηγήσω πώς συνεργαζόμαστε εμένα με τους ΔΕ. Και ε, κατακλείδαμε είναι εξή. Η Frontex, η Ευρωπαϊκή Συνορική και Εκτοφυλακή δεν είναι η μόνη. Ε, το μόνο μέλος αυτής της οικογένειας, αλλά έχουμε πέραν της υπηρεσίας Frontex, έχουμε την ακτοφυλακή. Θέλουμε λοιπόν ε, να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τα ε, επαρκή μέσα και πόρους για να μπορούμε να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Ευχαριστώ κύριε Λεζερή. Αρχίζει ο ε, πρώτος γύρος. Θα ακούσουμε τους προσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων και θα μπορέσετε στη συνέχεια να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο και θα ακολουθήσει η δεύτερος. Ο κύριος Λέναρς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεζερή, για την ε, συνεισφορά σας σήμερα στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από πλευράς Λαϊκού Κόμματος, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλεια των πολιτών, αποτελεσματικός έλεγχος και φύλαξη των συνόρων, για να μπορούν να κυκλοφορούν και ελεύθερα ε, οι άνθρωποι ε, στο εσωτερικό του χώρου Σέγγεν και να έχουν και εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, τεράστια ευθύνη. Και χάρηκα πολύ με τη νέα εντολή που σας δόθηκε και μεταξύ αυτών 10.000 ε, επιπλέον συνοριοφύλακες και λιμενικούς. Ε, πραγματικά τα έχουμε συζητήσει, αυτά τα είπατε κι εσείς εκτενώς και το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να είναι ενήμερο και να τηρείται ενήμερο για τα βήματα που λαμβάνονται ε, ως προς το νέο αυτό κανονισμό και την υλοποίησή του. Αναφερθήκατε στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να το μάθουμε κι εμείς για να ε, το κοιτάξουμε. Ε, δεύτερη ερώτηση και πάλι για την εφαρμογή πέρσι ολοκληρώσαμε ε, την αναθεώρηση του ΣΥΣ, του Σύστημα Πληροφόρησης Σέγγεν και χαρήκαμε πολύ που το καταφέραμε. Εδώ αφορά και το Frontex και τις ομάδες του και αυτό θα σημαίνει μεγάλη προσπάθεια για την εφαρμογή. Και εμείς επιμείναμε στο Κοινοβούλιο ε, σε μια αυστηρή προθεσμία για την ολοποίηση όλων αυτών. Τι θα γίνει με τη νέα ε, Frontex. Τρίτη και τελευταία ερώτηση. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων και φύλαξη ε, θα πρέπει να συμβαδίζει με την πλήρη, από ε, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Ε, είδαμε το καλοκαίρι τον Αύγουστο ένα ρεπορτάζ του γερμανικού καναλιού ARD και του Guardian όπου έλεγε ότι ο Frontex άφηνε κάποιους να κακομεταχειρίζονται τους μετανάστες. Ε, επίσης ε, για τα ε, σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο είδαμε ένα ρεπορτάζ από το Βελίο ότι δεν διαβιβάζεται στοιχεία στο front, από το Frontex. Παρακαλώ να μου απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Σίπελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Λεζερή. Ε, που μας δίνεται αυτή την επισκόπηση. Για να μην ειλικρινής, όταν διάβασα ε, τα έγγραφα για τη σημερινή συνεδρίαση, εξεπλάγει λίγο, διότι στην εισαγωγή έλεγε παρουσίαση ε, της αξιολόγησης τροτότητας. Ενδιαφέρον είναι αυτό, γιατί πήραμε μια επιστολή τον Ιούνιο με ένα έγγραφο που ήταν εμπιστευτικό και μας είπαν ότι προστατεύεται και με password. Δηλαδή σήμερα εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για όλες τις λεπτομέρειες ενός τέτοιου εγγράφου. Και αν επιτρέπετε, τότε γιατί προστατευότανε και έπρεπε να τηρήσουμε το απόρριτο και την εμπιστευτικότητα τότε. Και αν μισοεπιτρέπεται και μισοαπαγορεύεται, γιατί δεν συνεδριάζουμε και κλεισμένων των θυρών. Τι θα πει password protected document ε, για την ε, ευαλωτότητα, την τροτότητα. Ε, γιατί καμιά φορά εδώ στο Κοινοβούλιο κυκλοφορεί μια ιδέα για τα εξωτερικά μας σύνορα ότι θα πρέπει να ελέγχουμε όλους όσοι ε, περνούν τα σύνορα. Εμείς πάντα προειδοποιούσαμε γι' αυτό. Γιατί και στα εξωτερικά σύνορα καμιά φορά απλώς ο κόσμος περνάει τα σύνορα για να πάει για μπάνιο, ξέρω εγώ, ε, το Σάββατο ή να πάει στη λαϊκή ή ε, να πάει στο θέατρο. Τι θέλετε, να αλλάξουμε τη ζωή μας και τις ελευθερίες που είχαμε μέχρι τώρα. Σε ό,τι αφορά το σύστημα του ασύλου, ε, ε, αναφερθήκατε σε 10.000 επιστροφές, τις οποίες κάνατε προς χώρες. Έχετε ενημέρωση και σε ποιες χώρες πήγαν αυτοί, σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα ή πραγματικά στη χώρα ε, προέλευσης καταγωγής τους. Γιατί ε, επίσης είπατε ότι το προσωπικό σας θα οπλοφορεί ή οπλοφορεί. Οπλοφορεί παντού και πάντα. Και τι όπλα είναι αυτά που φέρουν. Έρευνα και διάσωση. Πολύ σύντομη ερώτηση. Έχουμε πολλές ιδιωτικές οργανώσεις που έχουν πρόβλημα να βρουν ασφαλή λιμένα. Τι γίνεται με το Frontex δεν άκουσα ποτέ να απαγορεύεται στο Frontex να καταπλέψει σε λιμάνι. Μπορείτε να μας το πείτε και ε, για τους 10.000 φύλακες που προβλέπονται. Αυτή θα είναι και της Frontex ε, υπάλληλοι, αλλά και αποσπασμένοι από τα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά ακούμε ότι δεν είναι εύκολο να βρεις προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο και με τα προσόντα που χρειάζεται. Ε, η Frontex αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα και πώς λειτουργούν όλα αυτά ε, για να δώσουν τα όσα υποσχέθηκαν όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τη Renew Europe, η κυρία Νετφέλτ. Παρακαλώ. Yes, thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. too. Um, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Λετζέρη. Ε, λεζερή. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις για την έρευνα και διάσωση. Εν συντομία, το ανέφερε ο συνάδελφος Λένατζε. Έχουμε αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ειδικέ επιχειρήσεις που δεν ε, ε, μιλάνε, δεν δίνουν τις πληροφορίες για την τοποθεσία και για την φύση του περιστατικού και των σκαφών που είναι σε κίνδυνο. Εμείς θεωρούμε πως πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πέρα από το ότι είναι ανήθικο και ε, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας επ' αυτού. Εάν για παράδειγμα επιχειρίες ε, μοιραστούν μαζί σας πληροφορίες, θα τις διαδώσετε κι εσείς και τι, ποια είναι η γνώμη σας για αυτή, την πρακτική. Έπειτα, διάφοροι ε, συνάδελφοι ανέφεραν πως οι δικές σας επιχειρήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα θρεμελιώδη δικαιώματα αλλά και με άλλους ευρωπαϊκούς νόμους όπως αυτόν για την διαφάνεια. Υπάρχει μια υπόθεση στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή όπου δύο άνθρωποι, δύο άτομα ή μάλλον δύο ΜΚΟ έχουν ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες για σκάφη που έχουν συμμετάσχει σε ε, αποστολή σε μια επιχείρηση και εσείς αρνηθήκατε την πρόσβαση με το επιχείρημα ότι ε, εσείς είστε μια υπηρεσία επιβολής του νόμου και δεν ισχύουν τα ίδια στάνταρ εφάνειας. Βέβαια είναι δύσκολο να πείτε τώρα κάτι γιατί είναι στα δικαστήρια υπόθεση, αλλά θα να καταλάβω. Γιατί πιστεύετε πως οι, οι κανονικοί, οι, κανόνες περί διαφάνειας δεν ισχύουν για το δικό σας οργανισμό. Και τέλος, όπως άκουσα και αναφέρθηκε ο κύριος Λένας, αναφέρθηκε σε μια άλλη υπόθεση όπου ο Frontex και οι υπηρεσίε του ε, έχουν ε, αναμειχθεί σε κακομεταχείριση ανθρώπων, στην Ουγγαρία επίσης. Θα ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις καταστάσεις, τι μέτρα λαμβάνετε και τι κάνετε για να προλάβετε τέτοιες, ε, τέτοια περιστατικά. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους η κυρία Στρίκα έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε για τις δραστηριότητε της Frontex. Οι κανόνες εξωτερικών συνόρων αφορούν βέβαια και την πρόσβαση στην προστασία και οι κανόνες του Σέγγεν και το κεκτημένο της Ένωσης. Εγώ... Έμαθα τις πρακτικές τις οποίες, και τις ερεύνησα τις πρακτικές που ασκείται στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στα εσωτερικά στην περιοχή Σέγγεν όπου γίνονται πολλές αποθήσεις πριν δηλαδή την διαδικασία ασύλου ε, επαναπροωθούνται προς άλλες χώρες και μάλιστα βία πολλές φορές. Επισκέφθηκα την ε, κρατική επικράτεια και τη βοσνιακή επικράτεια που γνωρίζετε πολύ καλά γιατί ο Frontex έχει και αποστολή, συνεργάζεται με τις συνοριακές αρχές και με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ακόμα και αν οι αθυρχές της Κροατίας αναγνωρίζουν πως ασκείται βία, ο Εθνικός Ομπουτσμαν της Κροατίας το αναγνώρισε, αλλά και ότι η Frontex επί τη βάση του συστήματος εξακολουθεί να λέει ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει και σε σχέση με τις εξελίξεις. Και αυτό με κάνει να με κατά πόσο ε, ε, λειτουργεί η, η λειτουργία παρακολούθησης της Frontex ε, ως οργανισμού. Πώς εξασφαλίζεται την ανεξάρτητη και σωστή παρακολούθηση των όσων γίνονται και το, της συμμόρφωσης που θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους ετούντες άσυλο σε εκείνη την περιοχή. Και επίσης θα ήθελα να θυμίσω ότι τουλάχιστον 40 επιπλέον ε, στοιχεία παρακολούθησης έχουν προβλεφθεί από το Ευρωκοινοβούλιο για να παρακολουθούν ε, τις ε, δραστηριότητες αυτές. Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Υπάρχουν και θα δούμε αν πρέπει να υπάρξουν και περισσότερα. τα καταρχάς να, δούμε, να υπάρχουν η δυνατότητα, αλλά να δούμε αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, ώστε να μας αναφέρουν τα σχετικά με τη συμμόρφωση. Ευχαριστώ, συνάδελφε, με την ε, παρέμβαση της κυρίας Τρίκ. Έχετε, έχετε Κλείνουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων των συντονιστών και τώρα μπορείτε να απαντήσετε για 10 λεπτά. Έχετε το λόγο, κύριε Λεζερή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις, τα διάφορα θέματα, διάφορες ερωτήσεις. Βοβλήθηκαν ερωτήσεις αρκετές για τα θεμελιώδη δικαιώματα, οπότε ίσως καλύτερα να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε η τηλεοπτική εκπομπή για υποτιθέμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων όπου ο οργανισμός ε, είχε υποτίθεται αναμειχθεί. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι τα όσα δημοσίευσαν τα μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου βασίζονταν σε 400 έγγραφα τα οποία αποκαλύφθηκαν από τον οργανισμό στο πλαίσιο μιας ε, αίτησης πρόσβασης, ε, δηλαδή μιας διαδικασίας πρόσβασης σε δημόσια σε έγγραφα δημόσιας υπηρεσίας. Ε, αυτό δείχνει πως είμαστε πλήρως σύμμορφοι προς την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Τι περιέχουν αυτά τα έγγραφα. Το γεγονός ότι εμείς σε κάποιες εκθέσεις λέμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου παίρνουμε τις πληροφορίες και μάλιστα από ΜΚΟ που λένε ότι άκουσαν για κακομεταχείριση ή για βία ή για παραβία, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλήσατε για την Ουγγαρία και για την Κροατία στις ερωτήσεις σας. πολύ συγκεκριμένα από τους 1.300 συνοριοφύλακες που έχουμε τώρα επιτόπου Έχουμε 8 στην Ουγγαρία που εργάζονται με βάρδιες και είναι, βρίσκονται σε ένα τμήμα των συνόρων που έχει μήκος 300 χιλιόμετρα. Αυτή είναι και η απάντησή μου. Πώς αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης ίσως με ορισμένα από τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα ή ε, τα θέματα νομιμότητας. Υπάρχουν θέματα συμμόρφωσης με, το, ε, ευρωπαϊκό, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάποιες φορές ε, βέβαια ο οργανισμός δεν μπορεί να αποφασίσει αν η εθνική νομοθεσία είναι σύμμορφη με την ευρωπαϊκή, γιατί αυτό είναι μακρά διαδικασία. Απλά να σας πω ότι στην Ουγγαρία έχουμε 8 συνοριοφύλακες. Στην Οκρατία δεν έχουμε επιχείρηση αναπτυγμένη εκεί στα, σύνορα, στα χερσαία σύνορα, ούτε στην κρατική πλευρά, ούτε στη βοσνιακή πλευρά. Πού και πού Έχουμε αεροπορική εποπτεία. Έχουμε δηλαδή αεροπλάνο που πετά στα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας στον κροατικό εναέριο χώρο, αλλά μέχρι στιγμής, και αυτή είναι η απάντηση του οργανισμού, ότι μέχρι στιγμής το αεροπλάνο αυτό ποτέ δεν έχει παρατηρήσει συγκεκριμένη ε, περιστατικό μεταχείριση. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι ανύπαρκτο, αλλά εάν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, πρέπει να είμαστε. Αυτή είναι η απάντηση του οργανισμού. Are so many reports about... Τώρα, γιατί γίνονται τόσες αναφορές για τα θεμελιώδη δικαιώματα που τις εκπονεί ο οργανισμός. Ακριβώς επειδή μας ε, ε, ε, μας απασχολεί το θέμα αυτό. Διαφορετικά δεν θα βρήκατε ποτέ εκθέσεις αναφορές που να μιλάνε για ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Το γεγονό ότι είμαστε διαφανεί και είμαστε απόλυτα σύμμορφοι με τη... τα ισχύοντα περί σε στα δημόσια έγγραφα, αυτό ε, αποδεικνύεται από το ότι δώσαμε στα μέσα που το ζήτησαν τα πληροφορίες που ζήτησαν τώρα. Γιατί ο οργανισμός αρνείται να αποκαλύψει κάποιες πληροφορίες, αρνήθηκε το 2017 ήταν, και αφορούσε την τοποθεσία σκαφών που επιχειρούσαν στην Κεντρική Μεσόγειο από την 1η Ιουλίου ή 1η Ιουνίου 2017 μέχρι τα τέλη του Αυγούστου 2017. Αρνηθήκαμε λοιπόν να δώσουμε αυτά τα στοιχεία διότι πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα επιβολής του νόμου. Όπως ανέφερα στην εισήγησή μου, ο οργανισμός μας και ο ρόλος μας είναι όλο ένα και πιο αναπτυγμένος. Ε, περιλαμβάνει και λειτουργίες ακτοφυλακής που σημαίνει επιβολή του νόμου στη θάλασσα. Ας πούμε το 2018 αναχαιτήσαμε 137 τόνους ναρκωτικών, τα οίμιση αυτών στη θάλασσα. Η καταπολέμηση λοιπόν της ε, ε, λαθρεμπορίας ναρκωτικών ή τις λαθρεμπορίας όπλων. Υπάρχουν ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις. Υπάρχουν διαφόρων ειδών διακινήσεις που γίνονται, εμπόρια και υπάρχει ανάγκη που, για συγκεκριμένους κανόνες που, θα, που ισχύουν για την αποκάλυψη τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών. Δεν λέω ότι δεν θα τα δώσουμε ποτέ τα στοιχεία, αλλά να γνωρίζετε και από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι, για παράδειγμα, η Frontex ω οργανισμό Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή, μαζί με το Europol και την Eurojust πρέπει να διέπονται από ιδιαίτερο νομικό καθεστώ όταν πρόκειται για το χειρισμό προσωπικών ε, στοιχείων και ευαίσθητων στοιχείων. Αυτό ισχύει για τι δραστηριότητε επιβολή του νόμου και όσον αφορά αυτήν ακριβώ τη δραστηριότητα ε, στη γη ή στη θάλασσα. Αυτή είναι η απάντηση. Το δικαστήριο θα αποφασίσει. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο διομεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί πως ε, πρόκειται περί χρηστής διαχείρισης. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Τώρα, για την ε, ανάπτυξη των 40 παρατηρητών για τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπεται από το νέο κανονισμό. Έχουμε ήδη αναπτύξει ε, επαφές με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γιατί στόχος μου είναι να συνεργαστούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα μας βοηθήσει να ορίσουμε καλύτερα τα προφίλ υπάρχει συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκούς οργανισμούς στον τομέα των ιστορικών υποθέσεων όπως είναι η Europol, η ΕΑΖΟ, η ΙΟΙΖΑ και θα θέλαμε να αναπτυχθεί τέτοια συνεργασία και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, εκείνοι έχουν τη γνώση, εμείς μπορούμε να μάθουμε από εκείνους και πρέπει να ενισχύσουμε τη λειτουργία της ε, παρακολούθησης. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αξιόπιστοι. Εφόσον συμφωνήσουμε ότι αυτή η λειτουργία θα πρέπει να αναπτυχθεί, θα πρέπει να γίνει με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Και τώρα μιλάμε για τη διαχείριση 40 παρατηρητών πρέπει να μιλήσουμε και για τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Για να σας δώσω μια εικόνα, ο προϋπολογισμός ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα πολλαπλασιάστηκε επί 11 υπό τη δική μου θητεία στον οργανισμό. Τώρα είναι 400.000 ευρώ ετησίως. Ήταν λιγότερο από 40.000 το έτος όταν εγώ ε, ε, διορίστηκα διευθυντής πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος, το, το, το γεγονός ότι όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο και με τον σωστό τρόπο. Και αυτό είναι κομμάτι της ε, εφαρμογής της νέας εντολής. Υπάρχει θέμα όσον αφορά το κλίδα κρυπτογράφησης και του κωδικούς. Ε, όπως σας είπα, δεν δημοσιεύονται αυτά γιατί έχουν πολύ ευαίσθητες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά στοιχεία, αλλά ε, για τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ε, χρησιμοποιηθούν λάθος σε εθνική συζήτηση ή θα μπορούσε επίσης να, να, να, να περιλάβει ε, εγκληματίες, τρομοκράτες ή οτιδήποτε. Τώρα, αναφέρθηκε επίσης στην κάμερα συνεδρίαση, σε δηλαδή κλεισμένο το θυρών, Πώς μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις ε, φυσιολογική, τη φυσιολογική υποχρέωση να αναφερόμαστε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να υπάρξει μία ε, κάλυψη της ανάγκης ε, προς αναφορά, αλλά και ταυτόχρονα προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών. Πάντοτε υπάρχει ανάγκη και πολύ Ευχαριστώ. θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ στο μέλλον ώστε να έχουμε μία συζήτηση που θα βασίζεται στο, ίσως στη μελλοντική έκθεση που θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο και να έχουμε μία κοινή συζήτηση αλλά και πιο εις βάθος, ε, καθώς αυτήν που ε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τον Ιούνιο, εσείς δεν ε, συνεδριάζατε. Το κοινοβούλιο δεν συνεδρίαζε. Τώρα για τη νέα εντολή και την ε, δημιουργία του μόνιμου σώματος, ο δικός χάρτης που ε, συμφωνήθηκε με την Κομισιόν. Ε, βεβαίως ανακοινώθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των καταρμέλων. Δεν το έχω φτιάξει εγώ, δεν μπορώ να σας το αναφέρω τώρα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα ε, δεν υπάρχει τίποτα εμπιστευτικό, αλλά είναι πολύ τεχνικής φύσης. Ε, να σας πω ότι αυτό είναι το λιγότερο, αυτό είναι, το χρονοδιάγραμμα ας πούμε, είναι αυτό που μας ζητά να εφαρμόσουμε η, ο αλλά είναι και ένα εργαλείο παρακολούθησης ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι ε, έχουν κάνει αυτό που τους αναλογούσε. Βεβαίως έχουμε ο καθένας τη δουλειά μας να κάνουμε, εμείς, η Κομισιόν, αλλά και τα κράτη-μέλη. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να ζητήσουμε ε, ε, ο καθένας να κάνει το μερτικό του από τον οδικό χάρτη. Τώρα, όταν πρόκειται για τους ε, αρμόδιος για την επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τώρα ξεκινάμε μια νέα εποχή όπου έχουμε βαδίζουμε σε βαθιά νερά και άγνωστα στην πρακτική της Ένωσης στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, αλλά δεν είναι άσχετο όσο αφορά την σύγκριση επιδόσεων και βεβαίως οι ε, επιδόσεις είναι των κατών μελών φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι να είμαστε το ίδιο πετατικοί με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή να είμαστε βέβαιοι πως υπάρχουν συγκεκριμένα τεστ, ψυχολογικά τεστ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τι είδους ε, όπλα, γιατί αυτά θα αναλυθούν σε αυτό το χρόνο. Ε, ε, τώρα, για τη γεωγραφική ισορροπία να πω ότι θέλω πάλι να ευχαριστήσω το Κοινοβουλίο που στήριξε τη διάταξη που πρότεινε η Κομισιόν για διαφορετική πληρωμή, ώστε να βληθεί ο κίνδυνος γεωγραφικής ε, μη ισορροπίας, έλλειψης ισορροπίας. Δυστυχώς ε, το Συμβούλιο ε, το απέρριψε αυτό και εάν δούμε ότι υπάρχει δυσκολία εξέβρεση γεωγραφική ισορροπία, θα το αναφέρω στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, στη Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Λεζερή. Σας ευχαριστούμε για την εξαντλητική σας απάντηση. Θα πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων τώρα. Είναι μακρύς ο κατάλογος ε, των βουλευτών που ζήτησαν το λόγο. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το ένα λεπτό που θα σας δώσω. Αλλιώ θα σα ε, κλείνω το μικρόφωνο. Ο κύριος Ράτεφ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λετζερή ε, για ε, την παρουσίαση που μας έκανε. Θέλω να σας πω όμως ε, ότι ακόμα αντιμετωπίζουμε τον απόϊχό της κρίσης του 2015. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά άνοιξε η Βαλκανική Οδός και είδαμε στα ελληνικά σύνορα τεράστια πίεση και μόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου περίπου 600 έφτασαν ε, στη Λέσβο ε, διαμέσου της Τουρκίας και οι περισσότεροι είναι Αφγανοί πολλοί φοβούνται μήπως επαναληφθεί η κρίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κύμα τον ασύλων. Θα πρέπει γρήγορα να κινητοποιηθεί ο ενισχυμένος Frontex. Ο Frontex εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ε, στην ε, φύλαξη των συνόρων. Και η δική μου χώρα, η Βουλγαρία, έχει ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Ρουίθ Ντεμπέσα. Σας ευχαριστώ κύριε Λεζέρη. Εδώ είμαι στα αριστερά σας. Ε, γεια σας. Ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ε, time. Ε, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να απαντήσετε. Μπορεί να το απαντήσατε παλαιότερα, αλλά επειδή είμαι νέο μέλος, το 2017 είχατε δηλώσει κάτι και σας παραθέτω, θα πρέπει να αποφύγουμε την υποστήριξη της διακίνησης ε, στη Λιβύη με το να έχουμε ευρωπαϊκά σκάφη να ε, σώζουν μετανάστες όσο γίνεται πιο κοντά στα λιβικά σύνορα ε, από κάτι άθλια σκάφη που δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηπλογιάσουν ούτε καύσιμα κτλ ε, τέλος παράθεση. Αυτό τι σημαίνει, ότι ΜΚΟ δεν θα πρέπει να συνεργάζονται εκεί στις αποστολές έρευνας και διάσωσης και θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ότι η Λιβική ακτοφυλακή μπορεί να αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Ο κύριος Πέτερς, ε, παρακαλώ. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ... Ε, εκτελεστική ε, διευθυντά, σα ευχαριστώ. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ στη Βαρσοβία το Frontex. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη. Έχω δύο ερωτήσεις, επαναλαμβάνω δύο και περιμένω σας παρακαλώ ε, απάντηση ε, για το προσωπικό, για τις προ, προσλήψεις. Ε, 10.000 μέχρι το 2027. Μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το 2024 που έχει αναφέρει ως ορίζοντα η κυρία Φόντερ Λάιεν όταν ε, φώνησε εδώ την παρθενική της ομιλία. Ε, και δεύτερη ερώτηση που επαναλαμβάνω. Ε, τα ευέλικα μέσα ενημέρωσης επανειλημμένα λέγουν ότι οι αξιωματούχοι της Frontex δεν διαβιβάζουν ε, σε σκάφη των μη κυβερνητικών οργανώσεων πληροφορίες από δικά σας σκάφη και αεροσκάφη σχετικά ε, με τους ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Και θυμίζω τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Για ποιο λόγο αρνείται η Frontex να διαβιβάσει ε, αυτές τις πληροφορίες σε παραπλέοντα σκάφη. Αυτό δεν παρεμβιάζει απλώς το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας, λέει η Πρόεδρος. Ε, η κυρία... Daily. Sorry, I didn't hear you calling my name. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα το όνομα μου. Κοιτάξτε, δεν απαντήσατε για τις αποθήσεις στα κροατικά σύνορα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν συγκρούσεις εκεί, βίες και το παραδέχτηκε και η πρόεδρος της Κροατίας. Και δεν απαντήσατε στο συνάδελφό μου. Και τι μας είπατε ότι δεν έχετε αρκετό κόσμο, μόνο 8 στα σύνορα της Ουγγαρίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε στελέχη, ότι δεν θέλετε να το αντιμετωπίσετε. Τα αεροπλάνα σας δεν βλέπουν τίποτα. Ε, δεν τα πιστεύω αυτά. Χιλιάδες ε, μαρτυρίες έχουμε ε, ανθρώπων των οποίων έχουν παραβεστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνατε τίποτα για να τα διερευνήσετε αυτά. Έχετε δημιουργήσει υπηρεσία παραπώνων και καταγγελιών. Αν δεν έχετε αρκετό κόσμο για να παρακολουθείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν έχω και πολύ τεράστια εμπιστοσύνη τώρα με βάση αυτά που μαθαίνω. Και τι κάνετε με την Ισραηλινή ε, κυβέρνηση, τον Ισραηλινό στρατό και τα Ισραηλινά drones, τα μη επανδρομένα. Είναι κρίμα, τώρα δεν έχουμε και χρόνο ομιλία στην Επιτροπή. Ε, ο κύριος Μπαρένα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λετζερή. Στα αγγλικά ο κύριος Μπαρένα. Δεν έχουμε χρόνο, θα μπω κατευθείαν στην ουσία. Το είπανε και άλλοι βουλευτές προηγουμένως. Σε μια συνέντευξή σας ε, στα μέσα ενημέρωσης επικρίνατε πολύ τις ΜΚΟ που σώζουν ζωές στη Μεσόγειο, στην έρευνα και διάσωση και κάποια στιγμή το είπατε έτσι ακροθυγός αλλά σαφώς ότι ορισμένες από αυτές τις ΜΚΟ συνδέονται, λέει, ε, με διακινητές. Ε, αυτό είναι γνώμη δική σας που ακούγεται περίεργη. Έχετε ακόμα αυτή την άποψη σχετικά με τα όσα συμβαίνουν κοντά στις Ιταλικές ακτές και έχετε στοιχεία για να το τεκμηριώσετε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά εγώ. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω σε ένα λεπτάκι. Έχω μια ερώτηση για την ασφάλεια. Γιατί συμφωνούμε εδώ στην Επιτροπή μας ότι η ασφάλεια οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και προσπαθούμε να το προασπίσουμε. Αλλά τα σκάφη του Frontex τώρα ε, δεν είναι πάρα πολύ παρόντα στην κεντρική Μεσόγειο. Δεν αναλαμβάνεται και ένα ρίσκο, ένα ρίσκο για την ασφάλεια, για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Τι γίνεται με τον έλεγχο των υδάτων εκεί στην Κεντρική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, του τελευταίου μήνε. Και δεύτερη ερώτηση, πολύ συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να δεσμευτείτε ότι όταν βρίσκουμε κάποια σκάφη που κινδυνεύουν στη θάλασσα και έχουμε αυτή την πληροφορία, δεν μπορούμε να το δημοσιεύουμε μέσω του συστηματος marsat EMARSAT-C. Και αν όχι, γιατί όχι. Ε, ε, για την ε, στελέχωση καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε τις προσλήψεις με τρόπο επαγγελματικό, αλλά πώς θα εξασφαλίσετε την ανεξαρτησία του Γραφείου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν είναι η συνήθις διαδικασία προσλήψεων για τους παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους υπολείπους υπαλλήλους. Και πώς θα, θα μπορούσατε να περιγράψετε τη συνεργασία με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Ευχαριστώ κύριος Ματζίντ.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 Όπως προαναφέρατε, συνεργάζεται η Frontex με κάποια κράτη για την εφαρμογή των επιστροφών σε τρίτες χώρες, ιδίως όταν οι σε διεθνούς προστασίας έχουν λάβει αρνητική απάντηση. Υπάρχουν όμως βαθιές ανησυχίες για το τι γίνεται σε χώρες όπως η Ουγγαρία, που οι αιτήσει παροχής ασύλου γίνονται με βάση την εθνική νομοθεσία ε, και θεωρούνται μη παραδεκτές αυτόματα. Τρεις περιπτώσεις τουλάχιστον είχαμε αιτήσει και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε νέα παιδιά, οικογένειες, νεαρές που μπορούσαν είτε να πάνε Σερβία είτε να τους χειρίσουν στο Αφγανιστάν ε, με πτήση της Frontex. Και η ερώτησή μου είναι τι μηχανισμούς μπορεί να εγκρίνει η Frontex για να μην επιβάλλονται οι αποφάσεις ε, επιστροφής που δεν συνάδουν με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας ευχαριστώ κυρία Σπούρεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αναφέρω ακριβώς την ίδια περίπτωση, δηλαδή την κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της ε, Πολωνίας, Τέρας Πολ, με βάση ε, τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και διαφόρων οργανώσεων ε, για πρόσφυγες και από την Τσετσενία. Υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι τους γυρίζουν πίσω χωρίς να μπορούν καν να αιτηθούν διεθνούς προστασίας. Η Frontex έχει αναλύσει την κατάσταση κατά την άποψή σας δικαιολογημένη, είναι δικαιολογημένη και νομικά αποδεκτή αυτή η κατάσταση, έχει γίνει εξολόγηση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Βυσνιεύσκα. Και με εσάς θα κλείσει και ο κατάλογος των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θετικές ε, βρίσκονται δράσεις της Frontex Καταλαβαίνω ότι έχετε να αντιμετωπίσετε στο έργο σας τεράστιες πιέσεις και οι φυλακές σίγουρα θα πρέπει να δείξουν μεγάλα ψυχικά αποθέματα και πολλή αντοχή εν γέννη. Θα επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός που πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι ε, πρέπει να δούμε πώς υποδέχεται η Ευρώπη τους παράτυπους μετανάστες εσείς τι θέλετε συνάδελφοι, θέλετε να έχουμε σύνορα σουρωτήρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να μπαίνει όπως θέλει και όποτε θέλει οποιοδήποτε. Σας υπενθυμίζω ότι η εμπορία ανθρώπων με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό δεν γίνεται λόγος ε, στη, στα ΜΜΕ, είναι κάτι που και ούτε και εσείς το αναφέρετε άλλωστε είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Υπάρχει, όπως και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Τι ε, διαστάσεις προσλαμβάνει το λαθρεμπόριο ανθρώπων ε, μέσω από τη Μεσόγειο. Thank you very much. I, ε, Και Κάνκο. 36% μόνο των παράτυπων μεταναστών επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής τους. Ε, οι υπόλοιποι που πάνε πέφτουν στην παγίδα της πορνείας, της εγκληματικότητας, της κακοποίησης. Αυτό δεν είναι σίγουρα κάτι ευκταίο. Αναθεωρήθηκε ο κανονισμός της Frontex, μας είπατε, όμως ενισχύθηκε η εντολή σας για τις επιστροφές. Νομίζω όχι. Ποια είναι η άποψή σας τι προσδοκίες έχετε, τι ελπίδες ε, τρέφετε ε, για τη βελτίωση της κατάστασης, διότι εδώ μιλάμε και για τα δικαιώματα, για προστασία πολλών ανθρώπων που ε, πραγματικά τους εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεζερή, για λόγους μερίσχιας διάταξης θα σας παρακαλέσω να μην υπερβείτε τα 6-7 λεπτά στην απάντησή σας. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένος για την ανταλλαγή προφορίας για ε, την έρευνα και διάσωση. Φέτος, ο οργανισμός μας διέσωσε 26.000 ανθρώπους στη θάλασσα. 15.000 ε, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ελλάδα και ε, Τουρκία, 1.500 στην κεντρική Μεσόγειο και οι υπόλοιποι ήταν μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Όταν πετούν τα δικά μας αεροσκάφη, και απαντώ εδώ και σε μια άλλη ερώτηση, για την αλλαγή στην κεντρική Μεσόγειο. Υπήρξε αλλαγή ε, και μειώθηκαν οι αφήξεις κατά 80%. Και εμείς ενισχύσαμε την εναέρια παρατήρηση ιδιαίτερα στην Κεντρική Μεσόγειο και εκεί ε, παρατηρούμε σκάφη σε κίνδυνο, μετανάστες σε κίνδυνο και όποτε γίνεται αυτό ε, το διαβιβάζουμε ε, στο MRCC, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης στη Θάλασσα. Με βάση το διεθνές δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι να το δίνουμε αυτό στα τοπικά MRCC δεν μπορούμε να τα διαβιβάζουμε άμεσα σε κάποιο άλλο σκάφος, είτε αυτό είναι εμπορικό, είτε είναι μήκυο, γιατί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα θα πρέπει να συντονίζονται για λόγους προφανείς, αλλιώς κινδυνεύουν ζωές. Ενδεχομένω. Έρχομαι τώρα στην απάντησή μου για το πώς θα αποφύγουμε να ε, προωθούμε ε, παράνομες επιστροφές ή αυτές που δεν συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και πάλι έγινε μια ερώτηση για τα χερσαία σύνορα. Θα πρέπει να επαναλάβω για ποιο λόγο στην Κροατία δεν έχουμε αναπτύξει ε, δυνάμεις. Δεν μας θέλει η κροατική κυβέρνηση. Δεν είναι ότι εγώ δεν έχω πόρους, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσω ότι εγώ δεν μπορώ να αναπτύξω κάπου επιχείρηση σε ένα κράτος μέλος αν δεν με θέλει το κράτος μέλος. Για τις επιστροφές, πρόσφατα είχαμε κάποιες επιφυλάξεις ε, το, για ένα περιστατικό, μια έγκυος που ε, επρόκειτο να επιστραφεί από την Ουγγαρία στο Αφγανιστάν. Παρόλο που δεν είναι στη δική μας εντολή, συζητήσαμε με τις αρμόδιες ε, ουγγρικές αρχές και αποφάσισα εγώ να σταματήσω αυτή την επιστροφή. Ένα γεγονός σας αναφέρω. Δεν ξέρω αν συνάδει, αν δεν συνάδει με την εντολή μου. Μπορεί και να μην συνάδει. Αλλά είχα την αίσθηση ότι η σωστή απόφαση ήταν να αποτραπεί αυτή η επιστροφή. Και έλαβα την απόφαση αυτή σε ό,τι αφορά την πρόσληψη 10.000 φυλάκων πριν το 2024, νομίζω, ε, ε, ξέρω ότι η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν το δήλωσε στο Κοινοβούλιο και το επανέλαβε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι στιγμής δεν είχα την ευκαιρία να ε, έχω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα και δεν έχω να σας πω τίποτα παραπάνω. Έγινε επίσης μια ερώτηση Ε, για τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη μας, πέρσι στην Κρήτη, ε, το δοκιμάσαμε. Είναι drones βέβαια για πολιτικούς σκοπούς, όχι στρατιωτικούς. Ήταν συνεργασία ε, ανάμεσα σε μία ευρωπαϊκή εταιρεία και μία μη ευρωπαϊκή εταιρεία. Ήταν κανονικός διαγωνισμός όμως και προμήθεια ε, ευρωπαϊκή. Ε, σε ό,τι αφορά τις περιπολίες, αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει τους εγκληματίες ε, τις περιπόλους μας κοντά στα λιβικά ύδατα. Το 2017, όπως είπατε, έγινε αυτό και τότε το θέμα ποιο ήταν. Υπήρξε αύξηση των πνιγμών και αύξηση των αφήξεων και τότε το 2017, 2017 επιμένω, ε, το καλοκαίρι η Ιταλική κυβέρνηση και τότε ήταν υπουργό ο κύριος Μινιέτη ε, θεώρησε ε, ότι υπήρχε ανάγκη ε, να προχωρήσουν σε ένα κώδικα διοντολογίας για τις ΜΚΟ. Γιατί πολλές φορές είχαν μη συντονισμένες προσπάθειες έρευνες και διάσωσης και μπορεί να κινδύνευαν ζωές. Επίση, σε ό,τι αφορά τη συλλογή στοιχείων, αποδεικτικών για ποινικέ ε, υποθέσεις. Δεν λέω ότι ήταν οι εγκληματίε ή ΜΚΟ, αλλά όταν ε, πιάνει ένα καράβι ή το σώζει και υπάρχουν ε, διακινητές ή εγκληματίες σε αυτό το σκάφο, χρειάζονται επαγγελματίε αστυνομικοί για να μπορέσουν ακριβώς να συλλάβουν και εκείνους που ενέχονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε, ότι οι παράτυποι μετανάστες ουσιαστικά είναι θύματα. Είναι τα θύματα των διακινητών και υπάρχουν και πολλές εγκληματικέ οργανώσεις στα πλαίσια ε, αυτά. Το 2018 ε, βοηθήσαμε να συλληφθούν ε, περίπου χίλιοι διακινητές λαθρέμποροι. Αυτή είναι η δραστηριότητά μας και πραγματικά είναι και τμήμα ε, της ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Ζητώ συγγνώμη για τις ερωτήσεις που δεν μπόρεσα να απαντήσω, αλλά δεν πρόλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις που θα πρέπει να επαναλάβω. Ο κύριος Λέναρς σας είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το νοδικό χάρτη, το χρονοδιάγραμμα, το συντομότερο για τις δραστηριότητε σας. Και το δεύτερο, εμείς έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε με έγγραφα ευαίσθητα, ε, διαβαθμισμένα. Έχουμε και κανόνες και θα σας παρακαλούσαμε ε, στο μέλλον να μας στέλνετε έγγραφα χωρίς να χρειάζεται password για να τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λετζέρη. sorry. Δεν θα απαντήσω. Α, θέλετε να πείτε κάτι πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το τελευταίο. Ένα λεπτάκι μόνο. Well, are indeed, uh, rules, uh... Ε, ναι, όντως υπάρχουν κανόνες που εφαρμόζονται. Σε αυτό είχαμε μια ανταλλαγή ε, ε, στάνταρ διαδικασίας λειτουργίας μεταξύ του οργανισμού και της Επιτροπής σας και την επόμενη φορά που θα έχουμε ευαίσθητα έγγραφα, όπως είναι η εξολόγηση τροτότητας, είναι το μόνο που έχω υπόψη μου, έτσι ευαίσθητο έγγραφο, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον οδικό χάρτη. Ούτε ευαίσθητο είναι, ούτε διαβαθμισμένο, ούτε απόρριτο. Ένα χρονοδιάγραμμα είναι ένα οδικό χάρτη. Κατά την άποψή μου, ε, μπορεί να σα διαβιβαστεί, αλλά για λόγου τυπικού θα πρέπει να διαβουλευτώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και σε ένα λεπτό θα περάσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη. Συγγνώμη, Πρόεδρε, λέει κύριο Ρουίθ Πρόεδρε, δεν απάντησε στη δική μου ερώτηση ο κύριος Λεζερή γραπτό θα σα απαντήσει. Μην ανησυχείτε, γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νετβέλτ, πρόεδρε. Ε, ε, ναι, κυρία Νετβέλτ. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έλεγα. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα, αλλά έχω και θέματα. Ε, σημαντικές ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. Εδώ πνίγεται ο κόσμος στη Μεσόγειο. Και έρχεται το αφεντικό της Frontex και μας, λέει, μας δίνει απαντήσεις για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ε, που και δεν είναι σαφής. Λέει, λέγεται μόνο με το κέντρο συντονισμού θαλάσσιας διάσωσης ε, μοιράζεστε τα στοιχεία. Γιατί τι γίνεται με τα παραπλέοντα σκάφη. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα στέλνετε μόνο στο MRCC και πρόκειται εδώ για ζωές που πρέπει να σωθούν. Όταν έχουμε επίγουσες περιπτώσεις, μπορούμε καμιά φορά και συμβαίνει να χρησιμοποιούμε το VHF, τον ασύρματο, ε, για τη διάδοση πληροφορίας και όποιον ακούει. Ο κανονικός διεύλος για να έχεις επιχειρησιακή απάντηση είναι να το διαβιβάσεις στις αρμόδιες αρχές που ε, είναι αρμόδιες για το συντονισμό της θαλάσσιας διάσωσης, το κέντρο συντονισμού. Αυτό προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Και όταν οι χώρες δηλώνουν ότι έχουν ε, μία ζώνη έρευνας και διάσωσης και όταν ο Διεθνής Οργανισμός ε, Ναυτιλίας να θεωρεί και να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη χώρα, η συγκεκριμένη αρχή δήλωσε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εμείς δεν μπορούμε αυτό να το ψηφίσουμε. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τον ασύρματο, ε, το VHF των σκαφών για να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε όποιον βρίσκεται στην ακρόαση εκείνη τη στιγμή. Αλλά ε, η κανονική διαδικασία είναι μέσω του MRCC, γιατί αυτοί έχουν τη δυνατότητα, έχουν την συνολική εικόνα, ξέρουν που είναι τα σκάφη, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και φέρουν και την ευθύνη του συντονισμού ε, των επιχειρήσεων διάσωσης. Και εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε από εκεί και πέρα και να δώσουμε και τα δικά μας σκάφη και, το, και τον ε, εξοπλισμό μπαίνουν αμέσα υπό τη διοίκηση του κέντρου ο, ο θαλάσσιας διάσωσης, αν είναι κοντά τα σκάφη μας. Ε, ή λέμε ότι ε, μπορεί και το αεροσκάφος μας να εργαστεί πάντα υπό την αιγίδα του MRCC που θεωρεί ότι είναι αρμόδιο. Ε, συνήθως αυτό γίνεται με τα ευρωπαϊκά κράτη, είτε την Ιταλία είτε τη Μάλτα. Θυμάμαι μια φορά ότι είχαμε μια επαφή με την Τινησία Κάποιες φωνές ακούγονται από το κρατήριο. Ε, θα, να του τα πείτε όταν βγείτε από την αίθουσα, δεν έχετε το λόγο. Εμείς δίνουμε πληροφορίες σε όλα τα κέντρα συντονισμού ε, θαλάσσιας διάσωσης και αυτό μπορεί να αφορά και ένα κέντρο στην Τρίπολη, το αρμόδιο λιβικό κέντρο. Με διαβεβαίωσαν ότι όλα αυτά είναι σύνομα και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια και πορεί που έχουν ε, δοθεί για να αναπτυχθεί αυτό το κέντρο συντονισμού στην Τρίπολη. Ελπίζω να κατανοείτε σε ποιο δίλημα βρίσκομαι και επιχειρησιακά. Όταν βλέπω ότι υπάρχει ένα σκάφος που είναι πολύ κοντά στη Λιβύη και μπορεί να διασωθεί από τη Λιβική ακτοφυλακή και από κανέναν άλλον. Εμείς συνεργαζόμαστε με κάθε κέντρο συντονισμού που μπορεί να αναλάβει την επιχειρησιακή απάντηση. Και όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, το θέμα είναι να σώσουμε ζωές. Και αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν άλλαξε ποτέ, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Λοιπόν, τελειώνει εδώ αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Ε, έχουμε πολύ φορτωμένη η ημερησία διάταξη και περιορισμένο χρόνο. Αν έχετε ερωτήσεις, να το βρείτε τον κύριο Λετζέρη, πιάστε τον τώρα που θα βγει από την αίθουσα. Bien, estimados colegas, vamos a pasar al punto... Να περάσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο δέκατο σημείο τη ημερήσια διάταξη, που είναι η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την ιδιότητα του παρατηρητή στην ομάδα χωρών κατά τη διαφθόρα Γκρέκο, του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα κάνει μια παρουσίαση. conocen όπως γνωρίζετε, έχει ε, καθεστώς παρατηρητή ε, η Ένωση. Πρόσφατα το απέκτησε σε αυτή την ε, ομάδα χωρών. Η συνεργασία μεταξύ της ομάδας Γκρέκο και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ μέχρι τώρα ήταν πολύ χρήσιμη, ιδίως στα ζητήματα που απτώνται του κράτους δικαίου. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι θετική η θεσμική ενίσχυση των σχέσεων των δύο πλευρών. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένω να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι έχουν γίνει ώστε να δεχθεί η Γκρέκο αυτή τη νέα μορφή ε, συνεργασίας και πώς ακριβώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή μας ε, ως παρατηρητών ε, στις εργασίες της ομάδας. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα που συμπεριέλαβε στην ημερήσια διάταξη το πολύ σημαντικό αυτό σημείο, δηλαδή τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομάδα χωρών κατά τη διαφθορά. Εδώ και χρόνια μα απασχολεί το ζήτημα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώ εξέφραζε την υποστήριξη του και στην Κομισιόν για να σημειωθεί πρόοδο στη συμμετοχή τη Ένωση στην ομάδα Γκρέκο, το Συμβούλιο τη Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται στι κοινέ αξίε, προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και πράγματι η Ένωση συνεργάζεται με το Συμβούλιο τη Ευρώπη επί τη βάση ενό μνημονίου συνεννόηση, το οποίο συνήφθη το 2007. Ωστόσο, εδώ και καιρό η ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς παρέμενε ένας από τους λίγους φορούς του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον οποίο δεν υπήρχε ένα επίσημο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι οι δύο οργανώσεις δεν είχαν τη δυνατότητα να συζητούν και να συνεργάζονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Υπήρξαν κάποιες εξελίξεις πράγματι ε, την Άνοιξη και στις αρχές του φετινού καλοκαιριού και με τα χαράς να σας αναφέρω τα σχετικά. Πρώτα απ' όλα, το Μάρτιο του 2019 ο Γενικό Γραμματέα ε, της ομάδας ε, Γκρέκο απέστειλε επιστολή στην τότε Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου προτείνοντας η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να εκτάσει το ενδεχόμενο λαμβάνει μέρο σε εργασίες της ομάδας Γκρέκο ω Και αυτό έδωσε μια νέα δυναμική στο όλο, στο όλο θέμα. Ήταν καλοδεχούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Προεδρία και από την Κομισιόν. Αυτή η πρόταση παραμένουμε και εμείς δεσμευμένοι στη συνεργασία με την Κρέκο και ελπίζουμε έτσι να έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Τι έγινε τώρα τον Ιούνιο. Το Συμβούλιο στο Σχηματισμό Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις ε, εξέφρασε την υποστήριξή του στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως παρατηρή στο έργο της Γκρέκο και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα σχετικά μέτρα. Η Κομισιόν, όπως ε, αναφέρεται στην επιστολή του πρώτου Προέδρου Τίμερμανς και του Επιτρόπου Αβραμόπουλου, με αποδέκτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στάλει από την Κομισιόν επίσημο αίτημα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο εκφράζεται ε, η πρόθεση της Ένωσης να ζητήσει καθώς παρατηρητή στην ομάδα Γκρέκο. Και η Κομισιόν ταυτόχρονα έκρινε μια πρόταση που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση όταν συζητηθεί αυτό το θέμα ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί ναι, μεν η Κομισιόν μπορεί να καταθέσει αίτημα ε, συμμετοχή ω παρατηρητή, αλλά οι χώρε που είναι μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη είναι αυτέ οι οποίε πρέπει να εγκρίνουν το εν λόγω αίτημα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου να μπορώ να σας ε, ενημερώσω κάτι που φαντάζομαι το γνωρίζετε βέβαια γιατί υπήρξε ευρεία προβολή στο πλατή κοινό και στα ΜΜΕ ότι είχε αίσιο πέραση κατά θέση αυτού του αιτήματο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 10 Ιουλίου αποφάσισε να κάνει δεκτή την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, εργασίε του Γκρέκ ως παρατηρητή. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να τονίσω τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι να εκφράσω και πάλι την υποστήριξη της Κομισιόν και την άποψη ότι θα ενισχυθεί με τη συμμετοχή αυτή της Ένωσης η συνεργασία μας στον τομέα της καταπολέμησης ε, του διεθνούς εγκλήματος και της διαφθάσης και της προστασίας του κράτους δικαίου. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το καθώς Η Ένωση θα καλείται να συμμετέχει στη συνεδριά της ομάδας Γκρέκο αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου ούτε θα υπόκειται σε αξιολογήσει τη Δεν θα υπάρξει κάποια οικονομική επίπτωση και η Ένωση δεν θα τοποθετείται επισήμως στη διαδικασία αξιολόγηση ατομικών χωρών. Τέλο, και αυτό θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα και με αυτό θα ολοκληρώσω και την παρέμβασή μου, όπως εξέφρασε και ο πρώτος αντιπρόεδρος μιλώντα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είπε τέλο πάντων, το αίτημα και η έγκριση του αιτήματο δεν αποκλείει μελλοντικέ εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ομάδας Γκρέκο. Ευχαριστώ. Sí, muchas gracias. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σέπαλα. Νοητήτω. Μισό λεπτάκι. No, ciertamente solo tenemos una solicitud de preguntas. Ναι, έχετε ζητήσει το λόγο ε, κυρία Κινίτσι. Και όποιος άλλος θέλει παρακαλώ να πει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα και μας είναι πολύ προσφυλές ε, το θέμα της καταπολόμησης ε, της διαφθοράς. Η προσχώρηση της Ένωσης σε αυτό το πρόγραμμα, ακόμα και ως μόνο παρατηρητή, είναι σημαντικό, <coughs> αλλά θεωρώ πως το μέλλον θα πρέπει να προσχωρήσει πλήρως στην ομάδα των κατών που μάχονται κατά της διαφθοράς. Ευχαριστώ για την εισήγηση, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Ακριβώς ε, εξετάζοντας ε, το ενδεχόμενο ε, της πλήρους συμμετοχής της Ένωσης, θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν σκοπεύει να επεξεργαστεί μια ειδική ε, ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της ε, διαφθοράς που θα εντοπίσει τους τομείς κινδύνου, τις απειλές και τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο θέμα της πρόληψης και ανα και, και, και της ε, αναμένοντας κάτι πιο μακροπρόθεσμο. Αν, συνεχί, αν προτίθεστε να συνεχίσετε την παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επειδή προβλέπεται δημοσίευση σχετική από πλευρά τη Κομισιόν ε, την έκθεση ε, ε, κατά της διαφθοράς που δημοσιεύεται που μας δίνει δηλαδή την εικόνα, το να έχουμε μια ειδική έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αυτό θα ήταν πιστεύω πολύ σημαντικό. Επίσης θέλω να δω αν παρακολουθείτε την εφαρμογή της οδηγίας PIF που ορίζει την παθητική και την ενεργή ε, διαφθορά. Ε, δηλαδή ε, και σε επίπεδο ένωσης, δηλαδή κάποια ενέργεια η οποία βλάπτει τα συμφέροντα της Ένωσης. Ε, θα πρέπει τους επόμενους μήνες ε, να δούμε αν και κατά πόσο τα κρατημέλη έχουν μεταγράψει και εφαρμόσει τα πιο σημαντικά στοιχεία της οδηγίας, όπως η παράγραφος 4, εδάφιο 4 της οδηγίας αυτής. Να δούμε δηλαδή που βρίσκεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της οδηγίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με τα ερωτήματα που υπέβαλε η συνάδελφος Κινίτσι Στις 23 Ιουλίου μάλιστα υπέβαλα ε, και ερώτηση προς την Επιτροπή ακριβώς για να μας πει συγκεκριμένα τι σκοπεύει να κάνει πέρα από τη συμμετοχή ως παρατηρητή στο Γκρέκο και τι κάνει συγκεκριμένα, ποια είναι τα μέτρα για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρώ και τονίζω ότι η προσχώρηση στο Γκρέκο έγινε πολύ καθυστερημένα σε σχέση με την ε, δέσμευση που ανέλαβε το 2014 και δεν ε, μπορώ, και θα πρέπει να δούμε ε, τη συσχέτιση ανάμεσα στον οργανωμένο έγκλημα και την επικράτει ολόκληρη της Ένωση που θα πρέπει να προσανατολίσει τις ενέργειες της Ένωσης ε, όσον αφορά την εξέλιξη ε, ε, του οργανωμένου εγκλήματο τύπου μαφίας. Σα ευχαριστώ κύριε Ροπέρτη, κυρία Φεράρα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Κρέκο είναι σημαντικό βήμα μπροστά και αυτό το είχαμε μάλιστα εκφράσει την σχετική επιθυμία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με την ευκαιρία μιας ε, έκθεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, για την οποία ήμουν εγώ εισηγήτρια. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη συμμετοχή ε, ως παρατηρητή της ε, Επιτροπής στο πλαίσιο του Γκρέκο, που σημαίνει συμμετοχή στις συνεδριάσεις ε, και πρόσβαση στα έγγραφα που συζητώνται, πέρα από αυτό, τι μέσα θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα θέσει σε εφαρμογή για να βελτιώσει την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κυρία Φεράρα Η κυρία Ντόμπρες. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, ε η διαφθορά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά θα πρέπει ε, να την πατάσουμε, αλλά για να την πατάξουμε θα πρέπει να τη βρούμε πρώτα. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. μπορεί να δείξει σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες Πού βρίσκεται ε, η διαφορά και πόσο αποτελεσματικά την πατάσουμε. Δυστυχώς, εγώ είμαι από την Ουγγαρία και η κυβέρνηση αυτό που κάνει στους τελευταίους μήνες είναι να συγκαλύπτει τη διαφθορά και δεν δημοσιεύει τα στοιχεία. Για ποιο λόγο άραγε. Είναι προφανής η απάντηση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια έκθεση που λέει ότι η Ουγγρική κυβέρνηση είναι πιο διαφθαρμένη από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ούτε αυτές οι εκθέσεις δεν μπορούν να δημοσιευθούν στην Ουγγαρία υπήρξαν προβλήματα διαφθοράς, τα οποία έγιναν γνωστά μόνο μετά τις εκλογές και ο κόσμος ψήφισε προηγουμένως χωρίς να τα γνωρίζει. Αν δεν κυκλοφορούν οι εκθέσεις, αν δεν δημοσιεύονται, ε, δεν έχει κανένα νόημα, ιδιαίτερα στις χώρες που χρειάζεται αυτό επιγόντως. Θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται. Θα παρακαλούσα αυτού του είδους οι εκθέσεις να δημοσιεύονται εγκαίρως ε, και δεν επιτρέπεται τα κράτη-μέλη να τα συγκαλύπτουν όλα αυτά ε, για ίδια συμφέροντα. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, τι κάνει η ίδια τους η κυβέρνηση, αν έχει προβλήματα διαφθοράς και αν τα πατάσει. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Ο κύριος Νέσκα, έχω μία σύντομη ερώτηση, λίγο ευρύτερη και έχει να κάνει με το νέο μέσο που προτείνεται, τους νέους μηχανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος δικαίου έχω την εξής λοιπόν ερώτηση. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο Γκρέκο για αυτές τις ε, εκθέσεις και την ε, πραγματογνωμοσύνη στο νέο πλαίσιο και τη ενίσχυση του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η κυρία Στρίκ, ε, ε, ε, συμφωνώ με την προηγούμενη ερώτηση, τον Γκρέκο. δεν είναι μόνο για την πάταξη της διαφθοράς, αλλά υπέρ κάθε προστασίας ακαιρεότητας και τονίζω την ακαιρεότητα. Και αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το καθεστώς του παρατηρητή για να βελτιώσουμε τους ίδιους τους κανόνες μας συμπεριφοράς και διοντολογίας για να διαφυλάσσουμε την αχαιρεότητά μας ε, ως αξιωματούχοι, πολιτικοί κτλ. Θα υπάρξουν αναφορές ε, περιοδικές από πλευράς Γκρέκο για τις δικές μας επιδόσεις, θα χρειαστούμε συμβουλές. Μήπως μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό και στο εσωτερικό μας, ε, όσο γίνεται καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Σας συμβουλεύω να απαντήσετε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα, γιατί θα ξαναρωτήσουν μετά οι συνάδελφοι. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστώ. Δεν θα κάνω ό,τι μπορώ. Βεβαίως, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις πολλών βουλευτών σχετικά με τη σημασία ε, όχι απλώς της ε, πάταξης της καταπολέμησης διαφθοράς, αλλά και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Συχνά συμβαδίζει η διαφθορά με το οργανωμένο έγκλημα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Και το οργανωμένο έγκλημα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την ίδια την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Αυξάνονται οι οργανώσεις αυτές του οργανωμένου εγκλήματος και αυτό κινδυνεύει αυτή η παραοικονομία και το έγκλημα να ε, μπει και στην πραγματική ε, οικονομία των κρατών μελών. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω εγώ. Εγώ μια απλή τμήματάρχηση είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα να σας απαντήσω. Ε, και στο προσεχές μέλλον θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε πολιτικές συζητήσεις για το μέλλον και τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλω να αποφύγω όμως να απαντήσω στις ερωτήσεις που μπορώ αυτή τη στιγμή. Πρώτον, για τη δημοσίευση των εκθέσεων Γκρέκο, αυτό είναι θέμα των κρατών ε, που κάθε φορά αξιολογεί η Γκρέκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα είναι υπέρ της διαφάνειας. Αλλά δεν είναι η δική μας υπόθεση, ούτε μας πέφτει λόγος. Ε, και δεν αλλάζει αυτό από το καθεστώς του παρατηρητή που αποκτήσαμε. Ε, ε, τα κράτη τα οποία αξιολογεί η ίδια η Γκρέκο μπορούν να αντιταχθούν ή όχι στην παραδοσιακή δημοσίευση. Για το κράτος δικαίου σας ευχαριστώ για τη σύνδεση που κάνατε και τις αναφορές σας στην ανακοίνωση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο. Είναι ένα πολύ σαφέ στοιχείο στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο κράτος δικαίου. Η εκλεγμένη πρόεδρος είναι βαθύτατα προσιλωμένη στην υλοποίηση αυτής της πρότασης που έγινε τον Ιούλιο, επαναλαμβάνω, και βεβαίως με χαρά να συνεργαστούμε για την εφαρμογή αυτών, αξιοποιώντας όλη την πραγματογνωμοσύνη και την εμπειρία ή θέτοντα την εμπειρία μας στη διάθεσή σας για τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Κάποιοι συνάδελφοι δεν ξέρω αν θέλουν να απαντήσουν τίποτα. ¿Alguno de ustedes quiere Έχουμε χρόνο αν θέλετε να κάνετε καμιά συμπληρωματική ερώτηση. Αν όχι, ευχαριστούμε την κυρία Σύπαλα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε να μας στείλετε πιο λεπτομερή ενημέρωση. Ε, όχι εσείς, κάποιοι ε, προϊστάμενοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μέσης διάταξης. που είναι προγραμματισμένο για τις 4. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να τεντωθείτε έτσι λίγο, να χαλαρώσετε, έχετε Καιρό για ένα μικρό διάλειμμα. Στις 4 θα τα ξαναπούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που είστε πάλι εδώ. Να συνεχίσουμε το επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Το σημείο 9. Έκθεση Επιτροπή σχετικά με την αποκοινού επανεξέταση της εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑ για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, TFTP. Ο κύριος Λοράν Μισελ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΧΟΜ, Διευθυντής Ασφαλείας, θα, είναι, θα μας κάνει αυτή την παρουσίαση. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα, λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 όταν ε, άρχισε να εκδίδει εντάλματα και συγκεκριμένα για διάφορες πληρωμές. Μέχρι το τέλη του 2019 στο SWIFT συγκεντρώνονταν όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά μηνύματα σε δύο σερβερ, ένα στη ΣΥΠΑ, ένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, την 1η Ιανουαρίου του 10 άρχισε να ισχύει δεύτερη αρχιτεκτονική με την ζώνη επεξεργασίας στη ΣΥΠΑ και τη ζώνη επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να υπάρχει συνέχεια στο TFTP, από αυτές τις νέες συνθήκες με τις δύο ζώνες επεξεργασίας θεωρεώθηκε αναγκαίο να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν εγκρίθηκε η πρώτη εκδοχή. Έτσι το καλοκαίρι του 2010 υπήρξε δεύτερη εκδοχή. Το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του 2 Ιουλίου του 10. και τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου του 10. να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μισελ και μετά θα κάνουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο κύριε Μισελ εκ μέρους της Επιτροπής. Thank you, Chair. Um, dear honorable members. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή μου να παρίσταμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής από την Νέα Σύνθεση. Θα σας παρουσιάσω τώρα την έκβαση της αναθεώρησης της Συμφωνίας ε, TFTP. Πρώτα απ' όλα όμως, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ξέρω ότι ορισμένοι ε, είστε εξοικειωμένοι ιδιαίτερα βλέπω γνωστά πρόσωπα, αλλά για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, καλό θα ήταν να σας κάνω καταρχάς μια ενημέρωση για αυτή τη συμφωνία, και πώς αυτή λειτουργεί και μετά να έρθω στην ουσία του θέματος. Ε, το τι FTP σημαίνει πρόγραμμα χρηματοδότησης, ε, πρόγραμμα συγγνώμη, παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ο στόχος είναι να εντοπίζονται οι τρομοκράτες ε, μέσω των οικονομικών τους συναλλαγών των τραπεζικών συναλλαγών. Η συμφωνία αυτή μεταξύ Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών ε, θέτει όρους και προϋποθέσεις καθώς και ασφαλιστικές δικλείδες για την ε, μεταφορά μεταβίβαση συγκεκριμένων οικονομικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η συμφωνία Επιτρέπει επίση στην Ένωση και στα κράτη-μέλη τη να επωφελούνται του παράματο αυτού. Μπορούν να ζητήσουν δηλαδή την αναζήτηση οικονομικών δεδομένων όταν θεωρούν ότι υπάρχει εύλογη υποψία για τρομοκρατική δραστηριότητα. Η συμφωνία του TFTP λειτουργεί ω εξή. Οι ΙΠΑ στέλνουν έτοιμα. Κατά, σε μηνύα βάση λίγο πολύ. Για όλα τα χρηματοοικονομικά μηνύματα σε σχέση με χώρες που έχουν υψηλό σχετικό κίνδυνο εμπλοκή στις τρομοκρατικές ενέργειες. Μετά από έτοιμα από την Europol, πάροχος διαβιβάζει μια δεσμέτρων στη βάση δεδομένων TFTP. Η βάση δεδομένων αυτή δεν είναι προσβάσιμη από το οικονομικό συνολικό αλλά μόνο ατομικά και αν υπάρχει συγκεκριμένη διασύνδεση με κάποια τρομοκρατική υπόθεση. Οπότε οι αναλυτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μόνο όταν κάνουν ατομική αναζήτηση στη βάση δεδομένων, συγκεκριμένα για κάποιο άτομο, για κάποια οργάνωση που έχει σύνδεση με τρομοκρατία ή με χρηματοδότηση τρομοκρατίας. σε όλες τις συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε κάνουμε το ίδιο πράγμα. Έτσι και τώρα έχουμε τον πάροχο, τον εγκεκριμένο ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί αν τεκμηριώνεται σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, με τρομοκρατική ενέργεια ή υποψία. Και μπορούμε να δούμε live στο διαδίκτυο τι αναζητήσεις γίνονται και να μπλοκάρουμε ενδεχόμενα τέτοιες έρευνες, αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει ε, επαρκής ε, ένδειξη ότι σχετίζεται πράγματι με την τρομοκρατία συγκεκριμένη αναζήτηση. Η συμφωνία TFTP περιλαμβάνει και κάποιες άλλες προϋποθέσεις και ως παραδείγματο χάρη κανόνες για την διακράτηση των δεδομένων, ασφάλεια δεδομένων, αίτηση πρόσβασης, επικύρωση. Και έτσι τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών ε, διασφαλίζουμε ότι είναι αντικείμενο νόμιμης ε, επεξεργασίας. Πού βρισκόμαστε τώρα. Από τότε που υπήρξε συμφωνία, το 2010, είναι η πέμπτη αξιολόγηση αυτή που έχει διεξαχθεί και καλύπτει την περίοδο 35 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30 Νοεμβρίου 2018. Αυτή η αναθεώρηση, η επανεξέταση έγινε καταρχάς στη Χάγη 15 Ιανουαρίου στα, στρατηγείο της, στα κεντρικά της Europol για να δούμε κατά πόσον ε, ε εκπληρεί τους όρους αυτής της συμφωνίας και έπειτα στο οικονομικό, στο οικονομικό τον είπα. Κοινέ είναι οι έρευνες, αλλά την αξιολόγηση την κάνει η Κομισιόν. Εγώ ήμουν επικεφαλής ομάδας ως Διευθυντής Ασφαλείας. Με συνάδευε συνάδελφος του κάθε δίπλα μου, ο συνάδελφο του κάθε δίπλα μου και δύο εκπρόσωποι από τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών. Ποια ήταν ε, τα αποτελέσματα αυτής της επανεξέταση. Ε, είναι ικανοποιημένη η ομάδα επανεξέταση σε ό,τι αφορά την τήρηση τη συμφωνία και των ασφαλιστικών δικλείδων και όρων και προποθέσεων. Η αναλογικότητα των διαβάσεων δεδομένων εκτιμάται με βάση την αξία που είχαν αυτά τα δεδομένα για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Είναι σαφές ότι είναι έγκαιρα, ακριβή και αξιόπιστα τα στοιχεία που παρέχει το TFTP για τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών και χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Το TFTP βοηθάει στην ε, αναζήτηση και τον εντοπισμό τρομοκρατών. Στην έκθεση περιλαμβάνονται διάφορα παραδείγματα, μπορείτε να τα δείτε, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία και την σπουδαιότητα της TFTP στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το TFTP ήταν πολύ χρήσιμο. Προχώρησαν χάρη σε αυτό συγκεκριμένες ε, έρευνες ε, για τρομοκρατικές ενέργειες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Παρακολουθείτε συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή με βάση αναζήτηση από το TFTP και ακολουθεί έρευνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. 17 Αυγούστου 2017, δηλαδή δύο χρόνια από τώρα. Στη Ράμπλα, στη Βαρκελόνη, έπεσε ένα αυτοκίνητο σε πεζούς και ποδηλάτες. Λίγα ώρα μετά, στο Καμπρίλς. Και μετά από αυτό, πέντε ιδιώτες με μαχαίρια επιτέθηκαν σε ανθρώπους που στον δρόμο. Ζητήθηκε η βοήθεια της Europol. Μέσα σε δύο ώρες δόθηκε θετική απάντηση και δόθηκαν 24 of those leads became the basis 24 ε, δέσμες ε, πληροφοριών, στοιχεία, πληροφορίες. Θα δείτε ότι η συμφωνία αυτή έχει προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια. Ε, δυστυχώς βέβαια γιατί έχουν αυξηθεί και τρομοκρατικές επιθέσεις τον τελευταίο καιρό. 402 αιτήματα κατέθεσαν τα κράτη-μέλη της Ένωσης και Europol στο πλαίσιο αυτής της περίοδου που κάλυψε έρευνα, ενώ είχαμε 192 στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Ε, Οι πληροφορίες λοιπόν αυτές ήταν πάνω από 82.000 σε σχέση με 11.600 περίπου της προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού. Τεράστια αύξηση των πληροφοριών που δόθηκαν στις αρχές ε, των κρατών μελών. Ποια είναι τα βασικά παρίσματα; Βεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο και μόνο για το σκοπό της καταπολέμησης τρομοκρατίας και της χρηματοδότησή της. Και αυτό είναι το δίκαιο Μετά από αίτημα της Europol. Αφού έχει διαπιστωθεί ότι είναι στοχευμένο το αίτημα και ότι υπάρχει ανάγκη τεκμηριωμένη για την ε, αναζήτηση των πληροφοριών αυτών. Αυτές οι πληροφορίες ότι FTP όπως είπα, μπορεί να τα επεξεργαστεί κανείς μόνο αν είναι ατομικό ε, το αίτημα και υπάρχει παρακολούθηση του καθενός στοιχείου στη βάση δεδομένων για να διαπιστωθεί ότι υπάρχει σύνδεση με την τρομοκρατία. Η έκθεση επιβεβαιώνει πως ο μηχανισμός ελέγχου λειτουργεί σωστά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αποτελεσματική συνεργασία σε ό,τι αφορά την παροχή ε, πρόσβαση στα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά διακράτηση δεδομένων. Επιβεβαιώθηκε από την έκθεση ότι όλα τα δεδομένα τα οποία δεν τα διακρατούν για να τα μελετήσουν, διαγράφονται μετά πέντε χρόνια. Βέβαια, υπήρξε ένα συμβάν που οδήγησε διακράτηση κάποιων δεδομένων πέραν αυτή τη χρονική περίοδου των πέντε ετών. Οι Αμερικανικές αρχέ. μας ενημέρωσαν συγκεκριμένα για αυτό το συμβάν και όταν έγινε και η αξιολόγηση στην Ουάσιγκτον μας το επανέλαβαν. Δεν υπήρξε πρόβαση, απλά έμενε στο ηλισμικό. Ήταν δηλαδή ανθρώπινο σφάλμα και αυτό διορθώθηκε. ανεξάρτητοι ελεγκτές το επιβεβαίωσαν. Ότι δηλαδή δεν έγινε αντικείμενο επεξεργασία στο δεδομένο το συγκεκριμένο και έχει διαγραφεί έκτοτε. Τώρα, περιθώρια περαιτέρω βελτίωση. Πρέπει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η χρησιμότητα των δεδομένων που λαμβάνονται. Για παράδειγμα, αν δείξει η εξολόγηση ότι τα δεδομένα μια συγκεκριμένη χώρα δεν δεν συνιστούν σημαντικές πληροφορίες για τις έρευνες, θα πρέπει να είναι πιο περιορισμένες λόγια δεδομένων από αυτή τη χώρα. Οι Αμερικανικέ Αρχέ επίση θα πρέπει να βελτιώσουν του μηχανισμού αναθεώρηση τη αναγκαιότητα ε, τη διακράτηση δεδομένων, τα οποία εξάγονται για ειδική έρευνα. Όταν γίνεται λοιπόν μια έρευνα, εξάγονται από τη βάση δεδομένων τα δεδομένα αυτά και θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναθεώρηση, η επανεξέτασή του και η διαγραφή του να λαμβάνει χώρα όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Μία από τι δυσκολίε είναι ότι, αν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή και διαφανή, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν ενημερώνεται παρκώ πάντοτε για το ότι έχει κλείσει μια υπόθεση. Οπότε, αν έχει μια πληροφορία και κάποια δεδομένα που έχει εξαγάγει και τα έχει στείλει στι Ισπανικέ Αρχέ, για παράδειγμα, όπω είπα πριν για τη Βαρκελόνη, όταν έχει ολοκληρωθεί η δίκη ε, και μπορούν να διαγραφούν αυτά τα στοιχεία δεν είναι απόλυτα σαφές για τις αρχές και αυτό πρέπει να, βελτιωθεί. Άρα πρέπει τα κράτη-μέλη να παρέχουν ε, feedback σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που απελαμβάνουν από τι Αμερικανικές Αρχές για να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν δύο πλευρές. Και όπως είπα και για τη διαγραφή των δεδομένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα. Εν κατακλείδη γίνονται συστάσεις για την βελτίωση της συμφωνίας ε, TFTP στην έκθεση αυτή. Επίσης σημειώνει ότι είναι διαφανή η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και ότι παραμένει σημαντική για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Και παραμένω στη σας για οποιοδήποτε ερωτήσεις. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μισελ. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων για τους συντονιστές. Νομίζω ότι ζήτησε το λόγο η κυρία Σίπελ εξ ονόματος των σοσιαλιστών και οι υπόλοιποι. Η κυρία Σίπελ έχει το λόγο. Συγγνώμη, Πρόεδρε, νομίζω ότι προηγείται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Λενάς, πρώτος. Maybe the EPP coordinator should start. Έλεγα ότι προηγείται το ΕΛΚ. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα. Είχατε ζητήσει το λόγο. Δεν ε, είχατε το όνομά σας. Ζητώ συγγνώμη. Δεν σας είχε σημειώσει η γραμματεία. Είναι πολύ ευγενή και έχει την καλοσύνη να σα αφήσει να μιλήσετε πρώτο, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Καλά, δεν πειράζει, να μιλήσω και μετά. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και ο τρόπος με τον οποίο μας εξηγείτε πώς λειτουργεί το TFTP και λειτουργεί πολύ καλά. Και ε, έχουμε πληροφορίες ε, εγκαίρως, αξιόπιστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να ε, πατάσετε η τρομοκρατία και να προσάγονται στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Είπατε για τη Βαρκελόνη ότι ζητήθηκε πληροφόρηση από τη Europol και απάντησε μέσα σε δύο ώρες. Αυτό είναι στάνταρτ. Το δύο, μιλήσατε για 400 ε, τόσες ε, αιτήσει. Δύο ώρες είναι μεγάλο διάστημα, μικρό, είναι στάνταρ. Πόσο χρόνο χρειάζεται κάθε φορά ε, για να απαντούν. Για ποιο λόγο ρωτώ διότι προσωπικά πιστεύω ότι για την ευρωπαϊκά και η πλευρά είναι περίεργο το σύστημα. Θυμάμαι μια φορά από την Ευρωπόλ μια διαφάνεια για το πώς λειτουργεί και ακόμα και η στοιχεία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καμιά φορά ένα κράτος μέλος πρέπει να το ζητήσει από την Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ από τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί βγάζουν τα δεδομένα, τα στέλνουν στην Ευρωπόλ και η Ευρωπόλ στα κράτη-μέλη στον 21ο αιώνα ε, δεν είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος συλλογής ε, κρίσιμων πληροφοριών. Στην Επιτροπή για την Τρομοκρατία είχαμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα TFTP και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νομοθετική πρόταση. δεν υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία στην αναθεώρηση που κάνετε τώρα για το TFTP με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να έχουμε και ένα δικό μας σύστημα για την Ένωση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Λέναρς. Τώρα η κυρία Σίπελ που είχατε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν θα επανέλθω στην όλη συζήτηση για το TFTP, αλλά θα προσπαθήσω να εστιάσω σε τέσσερις ερωτήσεις γιατί ξέρω ότι θέλουν και άλλοι να μιλήσουν. Ερώτηση πρώτη. Στη συμφωνία είναι ξεκάθαρο ότι δύο εκπρόσωποι των αρχών προστασίας δεδομένων θα πρέπει να συμμετέχουν στην αναθεώρηση που έχει συμβεί ήδη. Αλλά είδα μια εξήγηση που λέει ότι αυτοί οι εμπειρογνώμονε συμμετείχαν εξ ονόματος ευρωπαϊκή Επιτροπής και όχι υπό τις άλλε του επαγγελματικέ ιδιότητες. Αυτό τι σημαίνει. Ότι δεν επιτρέπεται να συζητήσουν για τις δικές τους απόψεις, αλλά όλα θα πρέπει να ε, ε, τα επικοινωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερη ερώτηση. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ο Ευρωπαίος επόπτης δεν έχει λάβει ε, όλες τις άδειες ασφαλείας, άρα δεν μπόρεσε να ε, εποπτεύσει όλες τις πηγές σε πραγματικό χρόνο. Ε, τότε εσείς πώς μπορείτε να ε, λέτε ότι λειτουργήσε σωστά ο μηχανισμός εποπτείας καθ' όλη τη διάρκεια της αναθεώρησης. Έρχομαι τώρα στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το εξή. Αξιολογώντας το αίτημα του άρθρου 4 του Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμάει τα μηνύματα στις περιφέρειες του κόσμου ε, που δεν ανταποκρίνονται στο TFTT και αυτό σημαίνει ότι θα ζητηθούν λιγότερα στοιχεία από τον πάροχο που ορίζεται. Μετά από εννέα χρόνια δηλαδή είναι δυνατό ε, να συλλέγονται τόσα πολλά δεδομένα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει ότι χρειάζεται πιο ειδική προσέγγιση, πιο στοχευμένη, ε, παρόλο που το λέει ήδη η συμφωνία. Ένα άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την εξόρυξη των δεδομένων, τα δεδομένα που έχουν εξόρυχθει. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα, θα πρέπει να αναθεωρήσει το μηχανισμό για την ανάγκη διακράτησης ε, εξοριγμένων εντό εισαγωγικών δεδομένων θα πρέπει να κρατούνται μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ειδική έρευνα και ανάκριση για την οποία ζητήθηκε να χρησιμοποιηθούν. Το άρθρο 6 παράγραφος 7 της Συμφωνίας δεν επιτρέπει όμως στην Ευρωπα... στις Ηνωμένες Πολιτείες να διακρατούν τα δεδομένα αυτά, πράγμα που κάνουν, εξακολουθούν να κάνουν μετά από 9 χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Ε, από την ομάδα Renew Europe, η κυρία Ενετφέλτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε εργαστεί σε αυτό το θέμα για αρκετό καιρό ορισμένοι από εμά και το γνωρίζουμε και εσείς γνωρίζετε τις επικρίσεις μας που παρέμειναν άθεκτες την τελευταία εννέα αιτία. Γιατί ποιο είναι το βασικό ζήτημα εδώ. Από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν hidden δεδομένα, bulk data, πράγμα παράνομο. Μαζικά. Και εκπλήσουμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ικανοποιημένη ότι εφαρμόζεται σωστά ε, η ε, συμφωνία και προχωρείται σε μια σειρά συστάσεις όμως για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ε, τότε πώς μπορεί να δηλώνεται ικανοποιημένη, δεν το καταλαβαίνω. Όπως είπε και η Μπίργκιτ Σίπελ, λέτε ότι ε, τα αιτήματα δεν είναι αρκετά στοχευμένα και συγκεκριμένα. Λένε ότι έχουμε μόνο ένα αίτημα το μήνα. Ναι, κάθε μήνα μου ζητάνε όλα τα δεδομένα. Ένα αίτημα είναι. Και αυτό είναι όμως ε, χήμα όλα τα στοιχεία μαζικά. Και γιατί τα διακρατούν αυτά μετά από 9 χρόνια. δεν ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όχι μόνο η συμφωνία, αλλά ούτε η εφαρμογή της. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Ε, μιλήσατε για τη δυνατότητα να μπλοκάρονται κάποιες αναζητήσεις ε, ε, σε πραγματικό χρόνο. Πόσο συχνά έχει συμβεί αυτό. Επίσης, ε, λέτε ότι το, το Υπουργείο Οικονομικών μας δίνει κάποια στοιχεία τώρα γιατί στην αρχή δεν μας έδινε τίποτα. Είστε ικανοποιημένοι ε, θεωρείτε ότι δεν σας δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Και τέλος, ε, η εποπτεία ε, της εφαρμογής συμφωνίας γίνεται μόνο με την κοινή αναθεώρηση ή υπάρχει και άλλος τρόπος. Από το κοινό όργανο εποπτείας της ευρωπό. Αν δεν θέλει ενείς άλλο συντονιστή στο λόγο, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε αυτό το πρώτο γύρο για να περάσουμε στον επόμενο. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις μία προς μία. Γιατί στα περίοδο που προβλέπετε για να απαντηθεί ένα ευρωπαϊκό αίτημα, Πάντοτε πρόκειται για δύο με τρεις ώρες. Όταν είναι επίγον το αίτημα, ε, επί τη βάση ενός τρομοκρατικού ε, συμβάντος. Ε, ένα κανονικό αίτημα παίρνει δύο-τρεις μέρες να απαντηθεί. Για το γεγονός ότι η Europol λειτουργεί ως κόμβος, ως hub, νομίζω ότι η εντολή της Europol είναι να λειτουργεί ως hub. Και επίσης είναι πολύ χρήσιμο ότι τα κράτη-μέλη κάνουν αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομικό ώστε να ε, δηληστούν κάποια στοιχεία. Και λειτουργεί έτσι ως ε, φίλτρο. Πιστεύουμε πως αυτό είναι θετικό και βέβαια δεν υπάρχει καθυστέρηση στοιχείων ε, από τη Europol σε επίγουσες υποθέσεις. για το ευρωπαϊκό TFTP. Δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω αυτό. Η επανεξέταση δεν, έδωσε, δεν έδειξε ανάγκη για ε, τέτοια σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα, αν ρωτήσετε την προσωπική μου γνώμη. Τώρα όμως όσον αφορά την Μελλοντική Επιτροπή και για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα τέτοιου τύπου, ε, αυτό θα πρέπει να το δει η επόμενη ε, Επιτροπή και ο επόμενος Επίτροπος που θα αναλάβει ε, αυτά τα θέματα. Από τεχνική άποψης δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη επί τη βάση της επανεξέτασης. Τώρα, για τα όσα ρώτησε η κυρία Σίπελ, για την ε, το θέμα της ε, ασφάλειας και την ε, άδεια από την ασφάλεια, αυτό είναι αλήθεια, ώστε να μπορεί κανείς να ερευνήσει και να παρακολουθήσει την έρευνα μέσα στο Υπουργείο Οικονομίας, χρειάζεσαι το υψηλότερο βαθμό ε, της ε, έγκρισης ε, όσον αφορά την ασφάλεια στις ΕΠΑ. Τώρα, στην περίοδο που κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, υπήρχαν επόπτες από τον πάροχο της υπηρεσίας που έκαναν αυτή την έρευνα και εκτιμούσαν την ασφάλεια. Υπήρχε δηλαδή έλεγχος και όταν χορηγήθηκε πρόσβαση σε έναν εκπρόσωπο της Κομισιόν μπόρεσε εξ να εξετάσει όλες τις έρευνες που ε, είχαν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εξέτασε δηλαδή όλες τις έρευνες κατά τη διάρκεια της περίοδου όπου δεν ήταν διαθέσιμος και επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες έγιναν σε συμφωνία με την ε, ε, σύμβαση. Υπήρχε δηλαδή ένα κενό κάποιων μηνών που δεν ήταν ε, ε, παρόν, αλλά που μπόρεσε εξ να ελέγξει. Συλλέγονται υπερβολικά πολλά στοιχεία. Αυτό είναι ο ρόλος μας και η συζήτηση με τους Αμερικανούς είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να εξασφαλίσουμε την αναλογικότητα. Και αυτό κάνουμε, γι' αυτό και δίδουμε κάποιες συστάσεις ε, ώστε να εργαστούν περισσότερο για να μειώσουν τον αριθμό των ε, στοιχείων, τον όγκο των στοιχείων που συλλέγονται. Αυτή είναι μία από τις συστάσεις μας. Τούτου λεχθέντος υπάρχουν κάποιες χώρες θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει το γιατί, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες, ε, όπως στοιχεία που συλλέγονται από την Νότια Αφρική, δίνω ένα οποιοδήποτε παράδειγμα τώρα, και έπειτα εξ υπάρχουν ε, ε, υπάρχει συζήτηση και αιτιολόγηση της επιλογής αυτής και μετά βλέπουμε ας πούμε ότι μπορεί να είναι κόμβος για χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας, κάποια χρήματα δηλαδή να περνάνε από αυτή τη χώρα. Αυτή είναι μια διαρκής διαδικασία. Μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε και καθημερινά να πούμε ποια θα είναι αυτή η χώρα, γιατί οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν διάφορες χώρες για να μεταφέρουν χρήματα και διάφορα δίκτυα. Οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς ευέλικτοι και να προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Για τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί, έχουμε κάνει μια σύσταση για διαγραφή αυτών όταν δεν είναι πια απαραίτητα για, ε, σκοπούς, ε, για τους σκοπούς της έρευνας. Ε, για αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ο αριθμός των στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την, στη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας και συχνά ο χειριστής των στοιχείων δεν ενημερώνεται για το ότι έχει κλείσει η υπόθεση. Οπότε Ε, η ενημέρωση μπορεί αυτή να γίνει αργότερα, γιατί μια δικαστική διαδικασία μπορεί να πάρει ε, πολύ χρόνο και άρα τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί διατηρούνται το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να γίνει η επεξεργασία τους. Για το ερώτημα του κυρίου, της κυρίας συγγνώμη, Interveld, υπάρχει φορά στοιχείων χίδιν, αλλά οι έρευνες γίνονται μόνο ατομικής βάσης. Δεν γίνεται ανάλυση των, στοιχείων χείριν. Είναι μόνο ανάλυση ανά περίπτωση. Νομίζω πως απάντησα έτσι και στις δύο για τις έρευνες που, που έχουν μπλοκαριστεί. Δεν έχουμε στατιστικές για αυτές, αλλά Συμβαίνει κάθε μήνα να υπάρχουν μια-δυο ε, έρευνες που μπλοκάρονται και μετά συνεχίζεται η συζήτηση με τους αναλυτές του ε, διαχείρισης για να δούμε γιατί μπλοκαρίστηκαν και τι πήγε λάθος. Κάποιες φορές ε, προσπαθούμε να δούμε γιατί η αιτιολόγηση μια συνεχιζόμενης έρευνας του FBI δεν είναι αρκετά σαφής και άρα ο αναλυτής επανέρχεται ε, και προσπαθεί να εξηγήσει και να βρει την έρευνα. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Συμβαίνει, έχει συμβεί μια δύο φορές, αλλά ποτέ δεν υπήρξε παραβίαση της συμφωνίας. Κάθε φορά που μπλοκαρίστηκε η έρευνα έχει ε, συνεχιστεί αργότερα και σύμφωνα με τη συμφωνία. Τώρα, ε, όσον αφορά το ETPS, έχουν ε, κάνει πρόσφατα μια έρευνα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση, αλλά είδαμε το σχέδιο αυτής και είδαμε πως είναι σύμμορφη με αυτά που έχουμε εμείς ε, βρει. Τώρα το EDPS θα πρέπει να εκδώσει την έκθεσή του. Πάντως είναι καλό, καλά τα αποτελέσματα που βρήκαμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ε, θέσουν ερωτήσεις οι υπόλοιποι βουλευτές. Έξι έχετε ζητήσει το λόγο. Ένα λεπτό έκαστος για να μπορέσουμε να ακούσουμε και απαντήσεις. Πρώτος, ε, ο κύριος Ράντεφ. Ράντεφ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, ε, συνάδελφοι. Καλησπέρα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μούσελ που μας υπέβαλε αυτή την έκθεση η οποία ε, αναφέρεται σε συμφωνία μεταξύ Ένωσης και ΕΙΠΑ ε, και την επεξεργασία μηνυμάτων οικονομικών συναλλαγών Γι' αυτό βοηθά όταν γίνονται έρευνες για τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Στην έκθεσή σας λέτε ότι θα εφαρμοστεί το γεωγραφικό κριτήριο στην αξιολόγηση των διαφόρων μηνυμάτων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα μόνα στοιχεία που ε, απεξεργάζονται εκεί είναι αυτά που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση αυτής και ότι η συμφωνία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ώστε να μπορούμε πραγματικά να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρικμό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την εισήγησή σας και λυπάμαι που έφτασα λίγο καθυστερημένα και έχασα την αρχή. Θα ήθελα κυρίως να ακούσω τι γίνεται με την πρόληψη, δηλαδή η συλλογή αυτών των στοιχείων και αυτή η μεταφορά στοιχείων έχουν, έχει επιτρέψει να προληφθούν ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτη και ποιες είναι οι σχετικές στατιστικές, γιατί είναι ένας αυτός από τους στόχους αυτής της συνεργασίας να προληφθούν όσο γίνεται οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ε, μάλιστα. Ο κύριος Γκάρνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο που ήδη ανέφερε η συνάδελφος Ιντεφελτ. Νομίζω πως γίνεται η χρήση των στοιχείων αλλά και δεν περιορίζεται όσο γίνεται περισσότερο εφόσον υπάρχει έτοιμα μήνα με το μήνα Πώς αυτό σημαίνει περιορισμό σε συγκεκριμένες απειλές. Εγώ νομίζω πως αυτό δεν ήταν ο αρχικός σκοπός του, του Κοινοβουλίου, ούτε έχει, είναι σύμμορφο προς την απόφαση του EFG ε, για τα στοιχεία, για την προστασία των δεδομένων. Εγώ βλέπω ότι εννέα χρόνια μετά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας δεν υπάρχει καν κανένα πρόγραμμα για ευρωπαϊκό ε, ε, TFTP. Και έπειτα ε, το 2010 λεγόταν ότι χάρη σε αυτήν τη νέα συμφωνία οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στη διόρθωση των στοιχείων τους. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί ποτέ από ό,τι κατάλαβα. και ο ενδιαφερόμενο ε, Ευρωπαίος πολίτης ποτέ δεν θα ενημερωθεί για το ότι τα στοιχεία του δόθηκαν στο TFTP. Είναι δυνατόν τελικά να έχει κανείς πρόσβαση να μπλοκάρει ή να διορθώσει τα στοιχεία. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό TFTP ακόμα και νέα χρόνια μετά και το Συμβούλιο είχε πει ότι αν πέντε χρόνια μετά την έναρξη αυτής της συμφωνίας έπρεπε να έχει θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ευρωπαϊκό FTP και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχη πρόταση. Ευχαριστώ και παρακαλώ έχετε το νου σας στο χρόνο. Κύριε Ντέιλι. Okay, thank you, Madam Chair. Is it you, you are... Εμένα, ευχαριστώ σε μένα η το λόγο. Μπρέιερ. Ναι, εγώ θα μιλήσω λίγο περισσότερο από ένα λεπτό γιατί εγώ έπρεπε να μιλήσω στον πρώτο γύρο των συντονιστών. Ε, σας ευχαριστώ πολύ γιατί εξετάσατε τις, στην πράξη το TFTP. Η, ερώτησή μου έχει να κάνει με το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των ε, μαζικών μεταφορών δεδομένων, το άρθρο 4. Μπορείτε να μας πείτε πόσες χώρες έχουν επηρεαστεί από τα αιτήματα αυτά και πόσες είναι ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερη μου ερώτηση αφορά τα στοιχεία τα οποία έχουν εξαχθεί και στα οποία έχει υπάρξει πρόσβαση. Η έκθεση σας λέει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα διατηρηθούν μόνο όσο είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη έρευνα. Άρα δηλαδή ότι χρησιμοποιούνται ακόμα και μετά τη λήξη μιας υπόθεσης, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται εκεί. Ερώτημά μου είναι, υπάρχει καμία νομική κάλυψη στις ΕΠΑ που απαιτεί από τις αρχές να διαγράφουν ε, τα δεδομένα FTP από τη στιγμή που έχει κλείσει μια υπόθεση ή από τη στιγμή που δεν χρειάζονται πια ακόμα και σε ανοιχτέ θέμα καθόλου. Υπάρχουν κανόνες για ενημέρωση του αρχείου ότι έκλεισε αυτή ή δεν υπάρχουν σχετικες νομοθεσιες για αυτό το θέμα καθόλου Υπάρχουν κανονες για ενημέρωση ε, του αρχείου ότι έκλεισε αυτή η υπόθεση, ας πούμε. Έπειτα, μπορείτε να μας πείτε για τον όγκο των στοιχείων που έχουν εξαχθεί και που είναι αποθηκευμένα αυτή τη στιγμή. Πόσα στοιχεία δηλαδή έχουν αυτή τη στιγμή η ΕΠΑ, αν έχετε τέτοιες στατιστικές. Τρίτη μου ερώτηση αφορά την υπόθεση ενός ατόμου που ζήτησε την επαλήθευση και είπατε ότι δεν έχει ελεγχθεί αν υπήρχε βάσιμος λόγος ότι συνδεόταν με την τρομοκρατία. Οπότε ανησυχώ αν αυτό το μέσο που υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις τρομοκρατίας όντως χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους υποθέσεις ε, που έχουν σχέση με τρομοκρατία ή όχι. Αυτό το εξετάσατε και μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι κάποιος ε, ε, επιβλέπει κατά πόσο υπάρχει σύνδεση με την τρομοκρατία. Και τέλος ε, θα απηχήσω την ερώτηση της κυρίας Ιντεβελ. Πώς μπορείτε να λέτε ότι είστε ικανοποιημένο ότι τηρείται σωστά η συμφωνία από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες υποθέσεις που προανέφερα, όπου δεν τηρείται σαφώς η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ και συγγνώμη κύριε Μπρέγκερ γιατί ε, δεν σας είχα σημειώσει σωστά στο, στον κατάλογο εδώ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εγώ είμαι καινούρια για αυτά τα θέματα, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους γιατί πιστεύω πως πρόκειται για ένα πολύ προβληματικό πρόγραμμα και συμφωνώ βεβαίως ότι αποτελεί μεταφορά χίδιν ε, στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών ε, τον είπα και το γεγονός ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση αργότερα και ότι μας διαβεβαιώνεται ότι θα, η έρευνα θα είναι όσο γίνεται πιο στενή ή όχι, αυτό δεν μπορεί να μας καθυσυχάσει γιατί πολλά από αυτά τα μέτρα που λέμε δεν είναι νομικώς δεσμευτικά στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης εποπτείας όπως τόνισε η διαμεσολαβήτρια στη δική της έρευνα που αναγκάστηκε να κλείσει γιατί δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από το Κοινοβούλιο να εξετάσει κατά πόσο ήταν αποδεκτό, αποδεκτή ε, η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με μια ξένη κυβέρνηση όταν η διαμεσολαβήτρια η ίδια δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ζήτησε και είπε ε, ότι οι διατάξεις τεχνικές, ε, αντίθετα με την ίδια τη συμφωνία, δεν ε, μελετήθηκαν ποτέ από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πότε λοιπόν το Κοινοβούλιο θα γνωρίσει τις τεχνικές προδιαγραφές. Η τελευταία έκθεση διαμεσολαβήτριας έχει εφαρμοστεί πλήρως. Η ΕΠΑ επιτέλους θα τεθούν στη δημοσίευση και εκπόνηση εγγράφων. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Κινίτση έχει το λόγο. Μάλιστα σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο που ήρθε και μας έκανε αυτή την εισήγηση για το σύστημα TFTP και θα ήθελα να ρωτήσω η δυνατότητα να μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, τις ροές ε, χρημάτων για είναι από σημαντικό μέσο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αλλά κυρίως να προλάβουμε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ε, θα ήθελα να κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια είναι τα αποτελέσματα και ποιες είναι οι δυσκολίες σε σχέση ακριβώς με την απόκτηση και διατήρηση των στοιχείων που προέκυψαν, ας πούμε, σε σχέση με το σύστημα μεταφορά χρημάτων ε, με το σύστημα το οποίο ορίζεται, ε, ονομάζεται ΑΒΑΛΑ και που θεωρείται πολύ σημαντικό ε, μέσο χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κυρίως σε σχέση με την αγορά και την διατήρηση στοιχείων ε, εν γέννη σε σχέση με την πρόληψη της τρομοκρατίας, αλλά πιο συγκεκριμένα ε, για αυτό το σύστημα μεταφοράς ε, εμβασμάτων που ανέφερα. Ευχαριστώ. Έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε παρακαλώ. Να είστε πολύ περιεκτικός και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Well, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι σε τρία λεπτά δεν μπορώ να απαντήσω σε λεπτομέρειες σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων που ήταν πολλές και λεπτομερείς. Κύριε Ράντεφ, πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες, όντω. ναι, το πιστεύω. Και απαντώ και στην κυρία Ντέιλι για την έλλειψη εποπτείας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για το TFTP. Σας θυμίζω ότι την πρώτη συμφωνία την είχατε απορρίψει, η λεγόμενη συμφωνία SWIFT ήταν αυτή. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναδιαπραγματεύτηκε τη συμφωνία αυτή και λόγω της δικής σας πίεσης προσθέσαμε τους επόπτες στη συμφωνία. Και για πρώτη φορά υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και ελέγχει, εποπτεύει ε, όλες τις ε, αναζητήσεις που κάνουν στο πρόγραμμα οι Αμερικανοί. Αυτό δεν υπήρχε στην πρώτη συμφωνία και είναι ασφαλιστική δικλίδα, όντως. Ελέγχουμε τη σύνδεση με την τρομοκρατία σε κάθε μία από τις αναζητήσεις. Είναι μεγάλη αλλαγή σε σχέση με αυτά που είχαμε διαπραγματευτεί στην αρχή και γνωρίζουμε ότι χάρη στη δουλειά σας έγινε. Ας μην αυτομαστεγωνόμαστε ότι δεν έχουμε εγγυήσεις και ασφαλιστικές ε, δικλείδες. Εσείς την προσθέσατε αυτή την εγγύηση την επιπλέον. Για να απαντήσω στην κυρία Μπρικμό στα γαλλικά. Ναι, έχουμε πολύ συγκεκριμένα και σαφή ε, ε παραδείγματα ε, τρομοκρατικών ενεργειών που αποσοβήθηκαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται η επίθεση και το TFTP ε, επιτρέπει να αποκαλυφθεί το δίκτυο και να εξαρθρωθεί. Το κάναμε αυτό και επίσης επιτρέπει να κάνουν κάποιες ε, συνδέσεις και ε, να ανακαλύψουν στοιχεία που η αστυνομία δεν μπόρεσε να κάνει στο παρελθόν. Σε σχέση με τον κύριο Κέρνα, ότι αυτά είναι χίδιν στοιχεία δεδομένα, bulk data, στη διαβίβαση γίνεται αυτό, αλλά υπό τον έλεγχο της ε, Ευρωπόλ. Διαβιβάζονται, αλλά στη συνέχεια δεν έχει πρόσβαση ε, συνολικά το Υπουργείο Οικονομικών, μόνο σε ατομική μεμονωμένη βάση. Ε, σε σχέση με ένα ευρωπαϊκό TFTP, επαναλαμβάνω κάτι που είπα και προηγουμένως, σας παραπέμπω μάλλον σε αυτό, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Πόσες είναι οι χώρες που ενέχονται, αυτή η πληροφορία είναι εμπιστευτική. Έχουμε κάποια παραδείγματα. Εμείς έχουμε δύο επόπτες προστασίας ε, δεδομένων και ξέρουμε ότι η δουλειά αυτή που γίνεται είναι αναλογική και γι' αυτό όταν μας λέτε γιατί είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι γενικά από τη συμφωνία ε, έχει φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και ε, πραγματικά αυξάνει χρόνο με το χρόνο, γιατί δυστυχώς αυξάνονται και οι απειλές όμως και οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Γενικώ είμαστε ικανοποιημένοι, πάντως υπάρχει χώρος για βελτίωση και βέβαια κάποια στοιχεία μπορούν να βελτιωθούν στι ΗΠΑ όπως τα εξοριγμένα αυτά δεδομένα. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να υποχρεώνει το Υπουργείο Οικονομικό να, να σβήνει αυτά τα στοιχεία. Ούτε νομοθεσία που να υποχρεώνει τις αστυνομικές αρχές να τα επιστρέφουν Τα στοιχεία ε, ή όταν κλείνει η υπόθεση στη δικαιοσύνη να συνεχίζει η ροή των πληροφοριών προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ε, ένα τελευταίο για, από ρώτησε η κυρία Κινίτσι ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι μία από τις δυσκολίες είναι ότι οι τρομοκράτες γνωρίζουν αυτό το πρόγραμμα ε, και προσέχουν, αλλά πάντα κάνουν λάθη ακόμα εξακολουθούν. Ε, αυτή είναι η προσθέμενη αξία. Οι πιο προηγμένες τώρα ε, τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ε, τα κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιούν συναλλαγές χέρι με χέρι, χωρίς να περνάνε από τράπεζες κτλ. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση πάντα για την, το να εμβάσει κανείς χρήματα ε, έχουν γίνει όλα αυτά ψηφιοποιημένα και ε, δυσκολεύουμε τη ζωή των τρομοκρατών και την πρόσβασή του σε ρευστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μισελ και ολοκληρώνουμε αυτό ε, το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο και τελευταίο για απόψη. Ανακοίνωση τη Επιτροπή προ το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο Κατευθυντήριε γραμμέ για τον κανονισμό σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός 2018-1807 καθορίζει ένα νομικό πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή όχι προσωπικού χαρακτήρα. Γιατί αυτά τα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στο νόμο περί δεδομένων, το GDPR δηλαδή. Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2019 έχει δημοσιοποιήσει μια κατευθυντήρια γραμμή που ξεκαθαρίζει έννοιε όπως είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεικτέ δέσμε δεδομένων κτλ. Το λόγο τώρα έχει κομισιόν και συγκεκριμένα και ο Σαχστανέ από τη γάμα δελτα Connect για 15 λεπτά το πολύ. Good afternoon, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο να κάνω αυτή την εισαγωγή και θέλω να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο που μας κάλεσε να έρθουμε να σα παρουσιάσουμε αυτή την ε, κατευθύνια γραμμή για ε, την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, τον κανονισμό αυτό και τον κανονισμό GDPR. Φυσικά είναι στο επίκεντρο ε, των νέων επιχειρησιακών μοντέλων και της ε, τεχνολογίας πληροφοριών τα δεδομένα, ρομποτική κτλ. Όλα αυτά απαιτούν ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά και πρέπει να εξασφαλίσει τα ελευθερία αυτών των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στον τομέα της ασφάλειας, αλλά να προστατεύσουμε και την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των ε, συμπολιτών μας, ε, που πρέπει να εμπιστεύονται την επεξεργασία των δεδομένων τους ε, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα θέλουμε και οι επιχειρήσεις να έχουν ασφάλεια δικαίου, να ξέρουν δηλαδή και τι κανόνες πρέπει να τηρούν. Εξού και το Ευρωκοινοβούλιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί τη προτάσει τη Κομισιόν για την ελεύθερη ροή των ε, δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα ζήτησε η Κομισιόν να διαμοσιεύει τέτοιου είδου στοιχεία για το πώ αλληλεπιδρούν τα δύο νομοθετήματα μεταξύ του. Αυτό για τα προσωπικά και αυτό για τα μη προσωπικά δεδομένα. Όπω λοιπόν ε, ίσω γνωρίζετε, η ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένας, ε, το αντικείμενο κανονισμού που άρχισε να ισχύει από τα τέλη Μαΐου με στόχο να δώσει ασφάλεια δικαίου σε επιχειρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων τους που είναι ε, μη προσωπικού χαρακτήρα επιχειρηματικά δεδομένα. Και αυτό σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας της Ένωσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη αυτές τις, ε, στην επεξεργασία και ταυτόχρονα θα ισχύουν οι βέλτιστε πρακτικές. Το άρθρο 8.3 ορίζει ότι μέχρι την 29η Μάη του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει καθευθυντήριες γραμμές για την σχέση μεταξύ αυτού του κανονισμού και του GDPR, ιδίω ό,τι αφορά τα μεικτά, τις μεικτές δέσμες δεδομένων, δηλαδή που συναποτελούνται από δεδομένα προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα, είναι κάτι που χρησιμοποιούν ε, κανονικά σε συνήθι βάση αυτές οι επιχειρήσεις. Είχαμε πολύ στενή συνεργασία ευθύ εξ αρχής για την εκπόνηση της κατευθυντήριας γραφτής γραμμής με τη γάμα Just εσωτερικά στην Κομισιόν αλλά και με τον επόπτη για την προστασία των δεδομένων που μας έδωσε και πολύ σημαντικό feedback Ποιο είναι ο στόχο, ποια είναι η ομάδα στόχος, επιχειρήσεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το GDPR και ε, την ελεύθερη ροή δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. δύο αυτούς τους κανονισμούς που παρέχουν ασφάλεια δικαίου, αναγκαίο και για τις επιχειρήσεις και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επομένω, η κατευθύνει αυτή γραμμή ε, και αποσκοπεί εξηγεί τα δύο διαφορετικά κόνσεπτ, δεδομένα προσωπικού και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, την αρχή της ελεύθερης διακίνησης και των δύο κατηγοριών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγόρευση της απέτηση εντοπισμού των δεδομένων και στους διακανονισμούς και τέλος φορητότητα δεδομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και την ρυθμιστική προσέγγιση που υιοθετούμε σε αυτόν τον κανονισμό. Όπως έλεγα λοιπόν, στην πράξη περισσότερες περιπτώσεις οι δέσμες δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα και προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα. Στην αρχή ο κανονισμός για, για τα μη προσωπικά δεδομένα ε, ορίζει ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή για να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με το GDPR. Αυτό τον κανονισμό που θα τον λέω FFD από εδώ και πέρα ξεκαθαρίζει όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος ε, κακής αλληλεπίδρασης ή αλληλεπικάλυψης των νομοθετημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για συμπληρωματικά μεταξύ του νομοθετήματα. Η κατευθυντήρια γραμμή βέβαια εξηγεί πιο αναλυτικά πώ θα εφαρμόζονται στην πράξη, πώ πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη αυτά τα δύο νομοθετήματα και ποιοι είναι οι κανόνε. Ειδικά για την αποφυγή της υπονόμευσης στην πράξη των, δεδομέ... των κανόνων των κανονισμών αυτών από τις επιχειρήσεις και έτσι ενισχύεται ο ρόλο των κανονισμών. Υπάρχουν και άλλοι τομεί αλληλεπίδραση μεταξύ της ελεύθερη ροή και του GDPR. Και αυτό είναι τυχή που τη βλέπουμε. Δηλαδή, πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν το γνωρίζουν αυτό. Ότι δηλαδή το GDPR ουσιαστικά προστατεύει την ελεύθερη ε, ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν κάναμε τι διαβουλεύσει με τι επιχειρήσει, διαπιστώσαμε ότι πολλέ φορέ δεν γνώριζαν την πτυχή αυτή. Και είναι πολύ καλό που έχουμε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή που το υπενθυμίζει. Γιατί είναι νομοθέτημα με στόχο την αρμόνιση ο GDPR. Ουσιαστικά εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασία σε όλη την Ένωση και αυτό επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προσπαθούμε να τονίσουμε στην κατευθυντήρια αυτή γραμμή είναι η απαγόρευση του, της απέτησης εντοπισμού δεδομένων, data localization. Δηλαδή, κάτι που αφορά κυρίως τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να δούμε τι ακόμη φραγμοί υπάρχουν στην ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, να προβούν σε απαραίτητε μεταρρυθμίσει για να αρθούν αυτέ οι απαιτήσει εντοπισμού δεδομένων. Όπω θα θυμάστε, έγινε πολλή λόγο όταν κατέθεσε αυτό το κανονισμό η Κομισιόν για την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά του ορισμού και δι τον ορισμό μη προσωπικό χαρακτήρα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση μα στην περίπτωση αυτή για τον ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οτιδήποτε δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Και αυτό βέβαια επιτρέπει μεγάλη ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο αφορά την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον. Ίσως να είμαι λίγο αφηρημένος, ίσως ένα παράδειγμα. Αν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη και άλλες πρόοδε τεχνολογία που θα επιτρέπουν την ανωνυμοποίηση δεδομένων που σήμερα θεωρούνται ανωνυμοποιημένα, άρα μη προσωπικά. Άρα αυτή η κατηγορία δεδομένων θα γίνουν πλέον μη ανώνυμα και άρα θα εμπέσουν στον κανονισμό GDPR. Θέλουμε ομαλή λοιπόν απρόσκοπτη μετάβαση από τον κανονισμό στον άλλο και την εξασφάλιση ταυτόχρονα για τις επιχειρήσεις ότι στοιχεία βιομηχανικά που έχουν κάνει τη ρομποτική θα είναι καλυμμένα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες δεδομένων που μας ε, απασχολούν ε, ψευδο, αν, ψευδονυμοποιημένα στοιχεία σε έρευνες για παράδειγμα ε, αφαιρούμε τα προσωπικά δεδομένα και αποκαθιστούμε αυτά τα δεδομένα από ένα σύμβολο ή με έναν αριθμό. Μένουν τα υπόλοιπα δεδομένα αλλά όχι τα προσωπικά αλλά ναι. υπάρχει δυνατότητα επαναταυτοποίηση. Ξεκολουθεί αυτό να θεωρείται όμω προσωπικό δεδομένο. Η ψευδονυμοποίηση δίνει τη δυνατότητα να ε, ταυτοποιείται κατά κάποιο τρόπο ένα άτομο, αλλά με τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, συσχέτιση, δύο διαφορετικών δεσμών δεδομένων, και δεσμών δεδομένων μπορούμε να τους ταυτοποιήσουμε και στην καθοδευτήρια γραμμή τα εξηγούμε όλα αυτά, ότι δηλαδή παρόλα αυτά αυτά τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά. Άρα εμπίπτουν στο GDPR. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην κατευθυντήρια γραμμή εξηγούμε ότι δεν υπάρχουν γκρίζε ζώνες πλέον χάρη σε αυτή την προσέγγιση με τον ορισμό των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και τον ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του GDPR. Μη προσωπικά δεδομένα και ο ορισμός. Μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις μελλοντικές ε, εξελίξεις. Κάποια στοιχεία για τα μη προσωπικά δεδομένα. Δεδομένα δηλαδή που αρχικά δεν μπορούν να οδηγήσουν στα αναγνώριση αυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή αρχικά που ήταν προσωπικά αρχικά και έπειτα ανωνυμοποιήθηκαν. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. καιρικέ συνθήκε, βιομηχανική, ε, βιομηχανικό μηχάνημα, ένα μηχάνισμα διαμόρφωση, ε, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, κάποια δεδομένα ή ομαδοποιημένα δεδομένα που δεν μπορεί κανείς να τα ε, αποδώσει κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Um, uh, για να υπάρχει ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή επειδή είναι θολή συχνά η γραμμή μεταξύ αυτών των δύο μορφών δεδομένων, πολλές φορές έχουμε τις μικτές δέσμες δεδομένων. Δηλαδή κάποια από τα δεδομένα είναι μη προσωπικού χαρακτήρα, αλλά όταν συνδεθούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες είναι δυνατή η ε, ταυτοποίηση και αυτές είναι και περισσότερε περιπτώσεις. Ε, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρήσει έχουν στη διάθεσή του μικτές δέσμε δεδομένων. Πάλι να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Φορολογικό μητρό μια εταιρεία. Μη προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη πλειονότητά του, αλλά κάτω-κάτω στον λογαριασμό θα ε, δείτε το όνομα του επικεφαλής ε, λογιστή που υπογράφει. Άρα βλέπετε ποιος είναι. Βλέπετε το όνομά του υπάρχουν διάφορα τέτοια ε, δεδομένα από χρηματοπιστωτικού οργανισμού, τράπεζε, εκεί που αναφέρονται πληροφορίε του πελάτη, κάποιε λεπτομέρειε μια συναλλαγή που οδηγούν τελικά στην ταυτοποίηση του ατόμου. Υπήρχαν πολλέ ε, ερωτήσει για την έννοια του άρρηκτα συνδεδεμένου, inextricably linked, που μπήκε στον κανονισμό για την ελεύθερη μη προσωπικών δεδομένων νομικός ορισμός δεν υπάρχει για το τι θα πει αυτό, άρρηκτα συνδεδεμένα. Εμείς προσπαθήσαμε να το καταδείξουμε με παραδείγματα για να είναι πιο κατανοητή έννοια αυτή. Παραδείγματο χάρη, όταν περιλαμβάνει δέσμη δεδομένων προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα, αν τα διαχωρίσουμε τα μένα από τα δε, λόγω της λύση της πληροφορικής ή αυτό θα είναι αδύνατον ή αυτό θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό για την ε, ε, ουσιαστικά διαχειρός ε, διάκριση των δύο μορφών δεδομένων. Έτσι προσπαθούμε τέλο πάντων να εξηγήσουμε τι σημαίνει τα συνδεδεμένα. Και κάτι άλλο σημαντικό που το επενθυμίζουμε στις επιχειρήσεις με την κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι δεν υπάρχει ή αδίποτε υποχρέωση διαχωρισμού των διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων. Δηλαδή, και τα δύο νομοθετήματα παρέχουν εξασφαλίσεις ε, στις ε, επιχειρήσεις ότι μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μεικτές δέσμες δεδομένων με την προπόθεση βεβαίως να τηρούν τις ε, διατάξεις των δύο κανονισμών. Και αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές αλληλεπίδρασης που επενθυμίζουμε. Δηλαδή, ο κανονισμό για την ελεύθερη ροή μη προσωπικών αφορά το σκέλο των μη προσωπικών δεδομένων με την επιφύλαξη της εφαρμογής του GDPR για το τμήμα εκείνο που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σύνολο των δεδομένων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ε, κομμάτι της ε, κατευθυντήριας αυτής γραμμής. Τέλος, φορητότητα. Είναι και αυτή μια αρχή την οποία εξηγούμε στην καθετήρια γραμμή και εξηγούμε τις διάφορες έννοιες, γιατί η φορητότητα διαφορετικός εννοείται στο GDPR και διαφορετικώς στον άλλο κανονισμό. Στο άρθρο 20 του GDPR γίνεται λόγος για δικαίωμα των φυσικών προσώπων να λαμβάνουν τα τα οποία έχουν δώσει έναν ελεκτή δεδομένων ή να διαβάζουν τα στοιχεία του έναν άλλον πάροχο υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη τώρα ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, δεν προβλέπεται δικαίωμα φορτότητας. Αυτός ο κανονισμός επιλέγει την αυτορύθμιση ως προσέγγιση και προτείνει για την Κομισιόν να διευκολύνει την δημιουργία κωδικών συμπεριφοράς διοντολογίας για τη φορητότητα κάποιων δεδομένων. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που πρέπει να φέρει σε πέρα σε αυτό το έργο και το έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε μια ομάδα εργασία με πάνω από 200 οργανώσει επιχειρήσεων και μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ε, και χρήστες. Ήταν κάθετο το κοινοβούλιο ότι πρέπει οι χρήστες να εκπροσωπούνται. Και τους έχουμε λοιπόν και αυτούς ε, από όλους τους κλάδους οικονομίας, μάλιστα. Οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και να προβάλλουν τις διεκδικήσεις τους σε ό,τι αφορά τη φορητότητα μεταξύ διαφόρων παρόχων υπηρεσιών και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και Πραγματικά ελπίζουμε να είναι χρήσιμες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις. Προωθούμε μέσω διαφόρων βημάτων συζήτηση στη βιομηχανία την κατευθυντήρια γραμμή για να εξηγήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επιχειρήσεις πώς μπορούν να, να ε, και από τους δύο δηλαδή και από το GDPR και από τον κανονισμό των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργούν ένα κοινό χώρο δεδομένων και από αυτό τον κοινό χώρο δεδομένων μπορούν να αποφεληθούν τα άλλα Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πριν να δώσω το λόγο σε όσους το ζήτησαν, θα ήθελα να σας ε, πω το εξής. Εγώ γεννήθηκα τον 20ο αιώνα. Είμαστε στον 21ο, ο Τα τεχνολογικά στοιχεία έχουν αλλάξει, αλλά τα δικαιώματα τα ανθρώπινα όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και της προστασίας αυτών. Κάθε φορά που μιλάω, που με ακούω να λέγει γίνεται λόγος για κώδικα διοντολογίας, αρχίζω και ε, αμφιβάλλω και μετά και τα, αυτά τα υβριδικά και χίδιν στοιχεία πάλι και αυτά με κάνουν ανησυχώ. Όλα όσα έχουμε διαβάσει σε αυτό το τομέα δεν ε, μπορώ να πω ότι με καθησυχάζουν. το αντίθετο και ε, λυπούμε, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα και όχι δικό σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σίπελ, σαν συντονίστρια των σοσιαλιστών και μετά στον κύριο Μπρέι. Ευχαριστώ. Έχει περάσει και η ώρα. Και ε, θα συνεχίσω στα γερμανικά. Είναι πιο εύκολο για μένα τέτοια ώρα. την παρακολούθησα αυτή τη συζήτηση ε, πολύ εντατικά για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που κατατέθηκαν το Μάιο και αν ε, πρόκειται να συνοψίσω τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη στοιχείων και δεδομένων. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει υποψία ότι θα μπορούσαν να είναι προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρούμε το GDPR. Άρα, βασικά πάντα, να <laughs> το πω έτσι κάπως τραβηγμένα. Ρωτώ, συμβαίνει αυτό όμως. Δηλαδή, ή σας λένε οι εταιρείε ότι καλά, αυτό δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα και δεν χρειάζεται να το σεβαστώ. Ε, και θα συμφωνούσα λοιπόν με την Πρόεδρο, χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες αντί για κατευθυντήρια γραμμή. Ε, γιατί πότε είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πότε δεν είναι. Πάντα αυτό είναι ανοιχτό για τη συζήτηση. Στο τέλο τη παρουσίαση, ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ξεκάθαρα ότι τώρα θα παρατηρήσουμε τι συμβαίνει, γιατί να δούμε τι γίνεται στην πρακτική. Ε, ακόμα και στην νομοθεσία, ε, συχνά περνάει πάρα πολύ χρόνο, ακόμα και όταν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μια νομοθεσία για να ισχύει κάτι σε ένα κράτο μέλο, και με τι κατευθυντήριες γραμμέ δεν φαντάζομαι να είναι διαφορετική η κατάσταση. Και συμφωνώ με την Πρόεδρο, το αργότερο στι αρχέ του επομένου έτου, καλό θα ήταν να καθίσουμε ξανά και να δούμε τον υποκείμενο κανονισμό και τις κατευθυντήριες γραμμές και ίσως ε, από εκεί και πέρα να έχουμε περισσότερο υλικό ε, για να εκτιμήσουμε πώς εφαρμόζεται ή που έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Κύριος Μπράιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά ε, την ε, συνένωση, τη συλλογή των στοιχείων για την ανομιμοποίηση. Πόσες μονάδες πρέπει να συνενώνονται έτσι ώστε να θεωρούνται ανώνυμα τα δεδομένα. Ας πούμε, σε ένα νοικοκυριό, ε, αν είναι η μονάδα το νοικοκυριό. Πόσα νοικοκυριά πρέπει να συγκεντρώσετε για να θεωρηθεί ότι είναι ανώνυμα αυτά τα δεδομένα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι αντίστοιχη. Η ανωνυμοποίηση των ε, διευθύνσεων IP. Ε, πόσα ψηφία χρειάζεται να βγουν από μια διεύθυνση, από ένα τέτοιο δεδομένο για να θεωρηθεί ότι είναι ανώνυμο. Μπορεί να γνωρίζετε ίσως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις ανακοίνωσε ε, ότι θα ψάχνει κεντρικά χρήστες κάποιες ιστοσελίδας και πραγματικά αυτά είναι ενισχυτικά. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια αυτά και τις ερωτήσεις σας. Ζητώ συγγνώμη που δεν κατάφερα να σας πείσω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ε, πραγματικά είναι εδώ για να σας καθησυχάσουν ε, και δεν προεξοφλούν καθόλου ε, την υλοποίηση των κανόνων για την προστασία δεδομένων. Είναι πάρα πολύ ισχυροί αυτοί οι κανόνες για το GDPR και οι κατευθυντήριες γραμμές ακριβώς γι' αυτό υπάρχει για να εξασφαλίσει την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με το GDPR και γι' αυτό την εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή έρχεται να συμπληρώσει αυτές τις δύο νομοθετικές ε, πράξεις όπου ήδη είναι πάρα πολύ ορισμένοι οι κανόνες. Η κατευθυντήρια γραμμή έρχεται να εξηγήσει ε, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα δύο νομοθετήματα. Οι δύο κανονισμοί, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Και σε περίπτωση αμφιβολίας εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός GDPR, ε, η οδηγία. Ο κανονισμός, ε, αν υπάρχει έστω και παραμικρή αμφιβολία όταν είναι μεικτό το σετ των δεδομένων και υπάρχει έστω και κάτι που είναι προσωπικού χαρακτήρα, βρίσκει εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, GDPR. Για οποιασδήποτε άλλες ε, λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια κατηγορία συγκεκριμένα παραδείγματα σε μια κατευθυντήρια γραμμή, ποιο θα είναι το κατόφλι για τη συγκέντρωση ή ε, κάποιο είδος προσωπικών δεδομένων όπως είναι οι διευθύνσει IP ε, υπολογιστών. Υπάρχει ένας μηχανισμός και όργανα Εθνικές Αρχές για την Προστασία Δεδομένων και Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας ακριβώς για να καθοδηγεί για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Η ομάδα εργασίας 29 έχει εκδώσει αντίστοιχη ε, οδηγία για την ανώνυμοποίηση και ψευδονυμοποίηση ε, που ισχύουν. Να προχωρήσουμε τώρα σε άλλες ειδικέ ανάγκες αυτό θα πρέπει να ε, συζητηθεί μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας ε, δεδομένων ε, και πάντα υπό την αιγίδα και την έγκριση του Ευρωπαϊκού.